Καλημέρα. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση. Όταν έχουμε όμως τον Υπουργό μαζί μας εδώ, θα πρέπει να περιμένουμε να υπάρχει ένα ικανό ακροατήριο. Καταρχήν έχουμε λοιπόν την έγκριση της ημέρησης διάταξης. Εάν δεν υπάρχει αντίρρηση, νομίζω ότι μπορεί να θεωρηθεί δεκτή. Έχω κάποιες ανακοινώσεις σύντομα. Η επόμενη μας συνεδρίαση καταρχήν θα είναι την Τρίτη το πρωί, 1η Φεβρουαρίου και θα κάνουμε ακροάσεις με διάφορους υποψηφίους για την Προεδρία των τριών Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών, εποπτικών καλύτερα αρχών. Περιμένουμε ακόμα την επιβεβαίωση ότι η συνεδρία στις 7 η Φεβρουαρίου, Δευτέρα πρωί, Δευτέρα Πόημα, θα είναι ακρόαση με τον Jean-Claude Trichet, ο οποίος προεδρεύει του ε, Ευρωπαϊκού Ταμείου Ρυθμιστών. Ήταν το απόγευμα της 7ης ε, Φεβρουαρίου. Επίσης, οι συντονιστές συμφώνησαν να κάνουμε μια έκτακτη συνεδρίαση την 5η 10 Φεβρουαρίου το πρωί και στη μέση διάταξη αυτή τη συνεδρίασης θα είναι η τροποποίηση των συνθηκών σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο προϋποθέτει ένα πολύ σφιχτό χρονοδιάγραμμα και θα συνενωθεί αυτό με θέματα τα οποία προβλεπόταν αρχικά να εξεταστούν την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου που θα χρησιμοποιηθεί όπως είπα για ακρόαση. Θα <clears throat> πληροφορηθούν τώρα οι συγητές και οι συντονιστές εν καιρό για τις λεπτομέρειες αυτές. Επίσης πρέπει να σας πω ότι ο πρόεδρος Φων Φαν Ρομπόι δέχτηκε να είναι παρόν στις 15 Μαρτίου ε, στη συνάντησή μας με τις Επιτροπές των Εθνικών Κοινοβουλίων για τα οικονομικά θέματα. Πάμε τώρα στο σημείο 3 που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ και τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας της Ουγγαρίας, ο οποίος θα μας δώσει μια σύντομη παρουσίαση και θα ακολουθήσει ανταλλαγή απόψεων. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ πέρα μαζί σας. Μόλις έχει ξεκινήσει η Ουγγρική Προεδρία ως Προεδρεύων του Συμβουλίου Οικονομικών και Ούγγρος και ως Ευρωβουλευτής εκτιμώ πάρα πολύ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εξορισμού ή βρίσκεται στην καρδιά της δημοκρατίας, οπότε νομίζω πως ε, εδώ είναι το σωστό μέρος και η σωστή στιγμή να συζητήσουμε κάποια σημαντικά και ζωτικά ζητήματα. Ήδη έχει ξεκινήσει διάλογος μεταξύ Συμβουλίου και Κομισιών Και θα ξεκινήσει και διάλογος μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και εξορισμού θα καταλήξουμε σε ένα τριμερή διάλογο. Οπότε Συμβούλιο, Κοινοβούλιο και Κομισιόν είναι από κοινού υπεύθυνοι για να ενισχύσουν την Ευρωζώνη και να αντιμετωπίσουν τα ζωτικά ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Να σας πω λίγο έτσι, τα βασικά της Ουγγρικής Προεδρίας όταν μιλάμε για οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Ε, εν ολίγης θα ήθελα να τονίσω την σημασία αυτών των ζητημάτων κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Βρίσκονται στην καρδιά της Προεδρίας μας, αυτού του εξαμήνου. Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα, παραδείγμα παραδείγματος χάρη αλλαγή της συνθήκης, οικονομική διακυβέρνηση, έξι νομοθετήματα, το ευρωπαϊκό εξάμεινο που θα ξεκινήσει τώρα και ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Όλα αυτά είναι ανοιχτά. Αυτά τα τέσσερα Ζηματικά ζητήματα σχετίζονται μεταξύ τους και πρέπει να τα λύσουμε ταυτόχρονα για να στείλουμε ένα μήνυμα στις διεθνείς χρηματαγορές και στους ψηφοφόρους μας ότι ναι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πράγματι έχουμε κοινή ευθύνη και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ είμαι έτοιμος να συνεργαστώ στενά μαζί σας ε, επί όλων των ζητημάτων που είναι ανοιχτά. Θα ήθελα να αναφέρω επιγραμματικά τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσουν το Συμβούλιο Κοφίν το εξάμεινο που έρχεται. Βεβαίως, έχουμε το νομοθετικό πακέτο περί οικονομικής διακυβέρνησης. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Όπως είπα, να είναι η πρώτη φορά που θα γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε επίσης ε, το πακέτο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και την εφαρμογή, η, τη διαμόρφωση του μόνιμου μηχανισμού κρίσης το λεγόμενο Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Πρέπει επίσης να δούμε τι θα γίνει με τους G20 και με εξωτερικές δραστηριότητες εν μεταξύ και θα καλύψουμε και κάποια πολύ σημαντικά φορολογικά ζητήματα με νομικές πρωτοβουλίες. Και βέβαια έχουμε και την αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου, το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα ζητήματα αυτά και να σκιαγραφίσω το χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση και τα έξι νομοθετήματα, όπως όλοι ξέρουμε, η σημασία της ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης έχει τονιστεί, υπογραμμιστεί από την κρίση, όλοι το επισημάνομαι αυτό. Αντικατοπτρίζεται αυτό στην έκθεση της Task Force που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και στις έξι νομοθετικές προτάσεις που δημοσίευσε η Κομισιόν. Η σημαντικότερη πρόκληση είναι στο πλαίσιο της Οι πιο σημαντικές προκλήσεις στο πλαίσιο αυτό είναι δημοσιονομική πειθαρχία, η οποία θα ενισχυθεί με το να δοθεί σημαντικότερο ρόλος στο δημόσιο χρέος, στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης και επίσης ζωτική σημασία έχει η ενίσχυση του εθνικού δημοσιονομικού πλαισίου των κρατών μελών. Um, Επίσης, μια προτεραιότητα κλειδί για την Ουγγρική Προεδρία είναι να καταλήξουμε σε μια συμφωνία εντός του Συμβουλίου για τις έξι νομοθετικές προτάσεις μέχρι το τέλος ή το πρώτο τρίμηνο του 2011 το αργότερο. Η Προεδρία είναι αποφασισμένη να διεξαγαγεί έντονες ε, επίσημε και άτυπε διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να καταλήξουμε σε μια τελική συμφωνία με εσάς, τον συνομοθέτη, το δυνατόν. Η Προεδρία λοιπόν σκοπεύει να τηρήσει το πιεσμένο αυτό χρονοδιάγραμμα, είναι πιεσμένο πρέπει να πω, που συμφωνήσαμε στο Συμβούλιο του Δεκεμβρίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Θα αυξηθεί έτσι η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία των οικονομικών πολιτικών μας. Όλοι γνωρίζουμε όμως πως όλα αυτά απαιτούν τεράστιες προσπάθειες από όλα τα κράτη-μέλη και επίσης από την πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ως αποτέλεσμα θα επωφεληθούν οι οικονομίες όλων μας από την υιοθέτηση και εφαρμογή αυτού του νέου πλαισίου που θα στείλει ισχυρά μηνύματα για τις δεσμεύσεις των κρατών μελών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς ισορροπημένη και διαρκή ανάπτυξη. Οπότε είναι ζωτική σημασία να καταλήξουμε καποριστικά οριστικά όσον αφορά την οικονομική διακυβέρνηση. Τώρα για το χρονοδιάγραμμα. Το Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο όρισε το χρονοδιάγραμμα. Θα γίνει αλλαγή της συνθήκης. Και έχουμε τις έξι νομοθετικές προτάσεις και μέχρι τέλος Μαρτίου θέλουμε να έχουμε συμφωνήσει σε όλα αυτά στο Συμβούλιο. Κατόπιν και εντωμεταξύ βεβαίως θα θέλαμε να έχουμε άτυπες συναντήσεις και επίσημες συναντήσεις ε, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικά με την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων. Και μέχρι τον Ιούνιο σκοπεύουμε να έχουμε οριστικοποιήσει και εγκρίνει τις νομοθετικές αυτές τις προτάσεις. Θα ήθελα τώρα να επισύρω την προσοχή σας στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Όπως ξέρετε, η εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου του 2011 θα δώσει μια διάσταση ex ante στον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι το οποίο σημαίνει πως θα είναι πιο έγκαιρη η κατεύθυνση των κρατών μελών. Οπότε, η Κομισιόν θα φροντίσει το πότε θα υποβάλλονται τα εθνικά προγράμματα σύγκλησης και μεταρρυθμίσεων με στόχο βεβαίως την εκπλήρωση των στόχων του 2020. Όλα αυτά τα στοιχεία της ε, σύλληψης αυτής είναι πάρα πολύ σημαντικά, δηλαδή τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και ο στόχος 2020. Όλα αυτά συνδέονται και στόχο έχουν να ενισχύσουν την οικονομική ανάπτυξη, να αυξήσουν την απασχόληση και ε, να αντιμετωπίσουμε τα οικονομικά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα. Τώρα, με βάση τις ε, συζητήσεις ε, με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδώσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να χαράξουν ανάλογα και την πολιτική του στα κράτη-μέλη, να εφαρμόσουν δηλαδή αυτά τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα. Τέλος, πρέπει να πω πω γνωμοδοτήσει και συστάσεις που θα υιοθετηθούν μετά από αξιολόγηση των προγραμμάτων θα ληφθούν υπόψη κατά την προετοιμασία των εθνικών προπολογισμών. Τώρα, όταν μιλάμε για την τελική επιτυχία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, πρέπει να πω πως το Συμβούλιο ΕΚΟΒΗΝ προβλέπεται να υιοθετήσει συμπεράσματα τον Φεβρουάριο για τις ε, μακροοικονομικές προκλήσεις και τις δημοσιονομικές προκλήσεις και θα υιοθετήσουμε μια γενικότερη έκθεση το Μάρτιο. Με βάση τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου, τα κράτη-μέλη θα προετοιμάσουν και θα υποβάλουν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα και τα προγράμματα σταθερότητας και σύγκλησης. Αυτό, αυτή είναι η ουσία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, δηλαδή να έχουμε συνολικά εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων και σύγκλησης. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν και τα κρατημέλη και η Κομισιόν καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να εργαστούν με γρήγορους ρυθμούς έτσι ώστε να μπορούν να εγκριθούν το Δεκέμβριο κατευθυντήριες γραμμές αναχώρα. Οπότε βλέπετε πως έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα που ενέκρινε το Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 2010. Τον Ιανουάριο το Συμβούλιο Κοφίνη ήδη έφυξε τα ζητήματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και είχαμε και την ετήσια έρευνα ανάπτυξης τον Ιανουάριο. Μέχρι το τέλος Μαρτίου το ΕΚΟΦΗΝ θα ετοιμάσει μια συνολική έκθεση. Επίσης μέχρι το τέλος Μαρτίου το Συμβούλιο θα ετοιμάσει τα συμπεράσματά του για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τον Απρίλιο ολόκληρη Ευρωπαϊκή, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τα εθνικά με τα αριθμιστικά τους προγράμματα έτοιμα και όλα αυτά θα καταλήξουν στους προπολογισμού των κρατών μελών. Και ελπίζουμε όλα αυτά να καταλήξουν στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων του 2020. Τώρα. Στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, τους κανονισμούς τους οικείους για τις χρηματοπιστωτικές ε, υπηρεσίες. Σε ό,τι αφορά την κρίση η οποία επεσυνεύει, έγινε σαφές ότι είναι απαραίτητο να έχουμε καλύτερη ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα. Αυτό είναι κατάφορο. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη εκκινήσει υπό τις προηγούμενες προεδρίες και εξάλλου κατά τη διάρκεια του επομένου εξαμήνου θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτή την πρόοδο και να διευκολύνουμε τη συζήτηση για τα πολλαπλά νέα θέματα που έχουν ανακύψει. Κατά τη διάρκεια της ε, Ουγγρικής Προεδρίας θα πρέπει να δώσετε πρέψα προσοχή στην συνεκτικότητα και στο σωρευτικό αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών. Όπως ξέρετε δημιουργείται μια νέα εποπτική αρχιτεκτονική στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρεις εποπτικές αρχές. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει ήδη από τον Ιανουάριο του 2011. Να προσθέσω απλώ ότι είναι μια προτεραιότητα και της Ουγγρικής Προεδρίας να επιτύχει ταχεία ε, έγκριση της οδηγίας Omnibus, Omnibus 2 και είναι πρόθεσή μας επίσης να τροποποιήσουμε και την οδηγία Solvency 2, Φεργιώτα 2 δηλαδή, και την, ε, όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα για τις ε, εποπτικές αρχές για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρα στο έργο τους. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών είναι απαραίτητο να μειωθεί ο συστημικός κίνδυνος και να υπάρξει αυξημένη διαφάνεια στις, χρηματο... στις χρηματαγορές. Η ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού τομέα θα πρέπει να καλύψει και την αγορά παραγωγών και τα, τη λειτουργία κεντρικών οίκων συμψηφισμού. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι απαραίτητο να εξετάσουμε είναι γενικά η αγορά αξιογράφων. Οι γυμνές πωλήσει και ορισμένες ε, μορφές ανταλλαγής υποχρεώσεων, ανταλλαγή ανταλλαγής αθέτησης υποχρεώσεων τα λεγόμενα credit swaps. Με τον τρόπο αυτό θα πρέπει να αποφευχθεί να συνεχιστούν ορισμένες ε, εσωτερικές πολιτικές στα κράτη-μέλη που έχουν οδηγήσει σε μια κατάσταση αβεβαιότητας. Δεν θέλουμε να αυξηθεί αυτή η αβεβαιότητα, αντίθετα θέλουμε να μειώσουμε το επίπεδο αβεβαιότητας το οποίο επικρατεί στο σύστημα μας σήμερα. κάποια ψήγματα θα μπορούσα να σας δώσω επίσης σε σχέση με τη θέση μας σε ό,τι αφορά τα φορολογικά ζητήματα. Η Ουγγρική Προεδρία στοχεύει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά ώστε να μειωθεί η τωρινή ανισότητα, η διαφορά μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της φορολογίας. Θα καταβληθούν προσπάθειες για να μπορέσουν να γίνουν διαπραγματεύσεις για την ε, επέκταση της εμβέλειας της οδηγίας για την αποτεμίευση, ώστε να υπάρξει πολιτική συνένεση στα θέματα αυτά. Για την απαραίτητη αυτή η πολιτική συνένεση, όπως κατανοείται όλοι. Επιπλέον, θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις για τη μεταρρύθμιση του, του πλαισίου για την ενεργειακή φορολογία. Το Συμβούλιο του Οκτωβρίου ζήτησε ήδη από το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να ξεκινήσει την ε, συζήτηση για την, ε, χρηματο, για την φορολογία του, του χρηματοπιστωτικού τομέα. Και έχουμε ήδη 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν κάποια μορφή τραπεζικής εισφοράς ή τραπεζικού τέλους. Αυτό σημαίνει ότι είναι έφορη η στιγμή για να μπορέσουμε να συζητήσουμε ευρύτερα το θέμα της φορολογίας στο χρηματοπιστωτικό τομέα απόλυτα προσιλωμένη στη συνέχιση των συζητήσεων αυτών σε υψηλό επίπεδο. Με στόχο να μπορέσουμε να θεσπίσουμε ορισμένε βασικές αρχές. Χρειαζόμαστε σε αυτό το στάδιο το πρώτο να έχουμε τις θεμελιώδεις αρχές και στη συνέχεια θα θέλαμε να μπορέσουμε να επιτύχουμε και μια συμφωνία. Τέλος, να στρέψω την προσοχή σας στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπω ξέρετε, η θέση εφαρμογή της Συνθήκης Λισαβόνα έχει τροποποιήσει και του κανόνε που διέπουν τον προϋπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταγραφή αυτών των αλλαγών και η εφαρμογή του στην νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι το απαραίτητο. Επομένω, η Προεδρία δεσμεύεται να συνεχίσει με στενή συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα όργανα να προχωρήσει στην έγκριση τη απαραίτητη νομοθεσία για την εφαρμογή τη συνθήκη της Και φυσικά μέσα στο γενικό το πλανητικό οικονομικό πλαίσιο γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι εταίροι και άλλοι παίκτες μέσα σε εισαγωγικά και υπάρχει και μια εξωτερική, μια παγκόσμια διάσταση που πρέπει να λάβει υπόψη η Προεδρία μας. Σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση έχουν γίνει πολλά σε αυτό το γενικό επίπεδο για να υπάρχει μια πιο συντονισμένη απάντηση στις προκλήσεις που προέρχονται από την οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Οι G20 έχουν αποδείξει να είναι ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό φόρουμ για να αντιμετωπίσει παγκόσμιες πτυχές οικονομικής διακυβέρνησης. Και ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκπροσωπηθεί πρεπόντος και θα συντονίσει σωστά τη θέση της με τους άλλους εταίρους. Αυτό ευνοείται και από την συνεργασία της Προεδρίας των G20 και της Ουγγρικής Προεδρίας. Και μια τελευταία πρόταση σε ό,τι αφορά την εξωτερική διάσταση. Παράλληλα με αυτά που γίνονται στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος και το Συμβούλιο Κοφίν στο πρώτο εξάμεινο του 2011 θα ξεκινήσει την προετοιμασία της θέσης του σε ό,τι αφορά τα μακροχρόνια θέματα χρηματοδότησης, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Είναι επιτάπτως λοιπόν η κλιματική αλλαγή και θέλουμε ήδη να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μιας κοινή θέση για τη μακροχρόνια χρηματοδότηση της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Αγαπητοί λοιπόν συνάδελφοι, αυτά είναι το ζουμί ούτως υπήν του προγράμματος της ε, Ουγγρικής Προεδρίας και θα ήθελα να κλείσω τη σύνομη αυτή ενακτήρια παρέμβαση, τονίζοντας και πάλι τα βασικά γεγονότα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε μια κοινή και σημαντική ευθύνη. Εγώ θα ήθελα να αναπτύξω μια πολύ καλή σχέση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε την εξέταση όλων των θεμάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, που όπως είπαμε προηγουμένως είναι αλληλένδετα και τα οποία κρεμούν σήμερα. Και αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας μένει μία ολόκληρη ώρα για ερωτήσεις. Παρακαλώ τους συναδέλφους ε, να μας πούνε αν έχουν κάνει μια ερώτηση για να κλείσει και έχουμε Ζαμοργκοζές, Γιώργιον Κλούτερ, Ούντε Μπόμαν, Λεον Κόγκ. And Ildiko Pellet Αυτά τα ονόματα έχουμε μέχρι στιγμής. Ποιος άλλος θέλει, κάντε μας ένα νεύμα. Anybody else? Mr. Langen, if you're going to wait. Κύριε Λάγκεν, αν θέλετε, καλύτερα να το πείτε τώρα, όχι αργότερα. Θα δώσω το λόγο σε δύο-τρεις συναδέρφους και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις σύντομες ε, ερωτήσεις παρακαλώ και σύντομες απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας, νομισματική και οικονομική. Κύριε Υπουργέ, καταρχήν σας συγχαίρω για το πρόγραμμα που μας ανακοινώσατε και ελπίζω να τηρηθεί. Πάση περιπτώσει όσον αφορά την δική μας ομάδα, εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να προχωρήσουν τα διάφορα θέματα. Αλλά για να προχωρήσουν τα θέματα θα πρέπει η Προεδρία να είναι αποφασισμένη, να παίξει το ρόλο της όχι απλώς να είναι ένα φερέφωνο του Συμβουλίου. Θα πρέπει να είναι μια, ένας φορέας αναζήτησης λύσης και διαλόγου. Και σας ερωτώ, τι μέθοδο θα εφαρμόσετε προκειμένου να προωθηθούν τα δύσκολα θέματα που έχουμε στο τραπέζι, έτσι ώστε για μερικά από αυτά να έχουμε κάποια αίσια κατάληξη ή δυνατόν μέσα στο εξάμεινο της Προεδρίασης. Ξέρετε ότι ο νομοθέτης αντιδρά αργά σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές, πολύ αργά. Πρέπει λοιπόν να κινηθούμε γρήγορα, αλλά και όσο πιο καλά γίνεται, έτσι ώστε ως κοινοβούλιο να ληφθεί υπόψη και η δική μας θέση και άποψη. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, συνεχίζω με τη σειρά που έγραψα τα ονόματα. κύριος Κλούτερ, Γιώργιον Κλούτερ. Ευχαριστώ. Έχω ένα ερώτημα το οποίο αναφέρεται στην οικονομική διακυβέρνηση. Είδαμε τους τελευταίους μήνες, το τελευταίο έτος, μία σειρά μικρών χωρών ε, στον νότο της Ευρώπης, ε, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη έγιναν θύματα της κερδοσκοπίας, ε, κάτι το οποίο συνεισέφερε και στην χρέωσή τους. Οι προτάσεις οικονομικής διακυβέρνησης της Κομισιόν προβλέπουν τιμωρία των χωρών που δεν τηρούν τα κριτήρια υπερχρέωσης, αλλά εάν τουλάχιστον ένα μέρος των χρεών των χωρών αυτών δεν είναι δική τους ευθύνη αλλά αποτέλεσμα κερδοσκοπίας, τι άποψη έχετε για τις προτάσεις αυτές τιμωρίας, είναι αποδεκτό αυτό, από τη δική σκοπιά. Από τη δική μας ε, σκοπιά των αριστερών στο Κοινοβούλιο δεν είναι αποδεκτό, είναι αυτοματισμός και προς λάθος κατεύθυνση. Γιατί επιδεινώνει την κατάσταση των χωρών που προσπαθούν να βγουν από την κατάσταση στην οποία είναι. Μια δεύτερη πτυχή ανέφερα τους μηχανισμούς ε, που συζητούνται αυτή τη στιγμή από την Κομισιόν, οι οποίοι θα μπορούσαν στη χειρότερη των περιπτώσεων να επιδεινώσουν τα προβλήματα των μικρότερων αυτών χωρών. Πέρσι δε ΔΕΗ Κομισιόν στην ανακοίνωσή της ε, στις 16 Δεκεμβρίου για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού είπε πως στο μέλλον θα πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση κοινωνικών επιπτώσεων για όλα τα μέτρα τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Πώς το βλέπετε εσείς αυτό, δηλαδή αυτά τα οποία προτείνονται ως μέτρα εξοικονόμησης ε, θα αντέξουν σε μια τέτοια αξιολόγηση κοινωνικών επιπτώσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα. Και επιτρέψτε μου να απαντήσω στη σειρά που τέθηκαν. Καταρχήν στο ερώτημα του Ζων Πολ Γκοζές. Σας ευχαριστώ που, συζητείτε, που συνεχίζετε έτσι με το ερώτημά σας τα προηγούμενα, τις προηγούμενες συζητήσεις μας. Όπως είναι γνωστό, δεν είμαστε εκπρόσωποι άλλων φορέων εκτός από το παρόν και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι προτεραιότητες που έχουν διατυπωθεί από την Ουγγρική Προεδρία έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν την τωρινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στοχεύουν στο να κερδίσουμε το στοίχημα του μέλλοντος. Ως Ούγγροι είμαστε δεσμευμένοι να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να έχουμε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η ζώνη του ευρώ και να έχουμε ένα ισχυρό και ανθεκτικό ευρώ. Και όπως τονίσατε, και νομίζω πολύ σωστά, πρέπει να δείξουμε οκίτητα στην αντιμετώπιση αυτή, αλλά πρέπει να λάβουμε και τις σωστές αποφάσεις. Και η ταχύτητα λοιπόν, αλλά και η σωστή αντιμετώπιση είναι κεφαλαιώδης. Σε σχέση τώρα με την τεχνολογία που θέλουμε να εφαρμόσουμε. θα σας πενθυμίσω αυτά που είπε ένας γνωστός ιστορικός, ο οποίος είπε είχαμε τρεις κύριους πυλώνες ανάπτυξης στην ε, ιστορία της ανθρωπότητας, την κουλτούρα, την γεωγραφική θέση και τρίτον την ύπαρξη τεχνολογίας. Τα τρία αυτά στοιχεία λοιπόν συμβαδίζουν, πρέπει να συμβαδίζουν για να μπορέσει κανείς να έχει μια σημαντική πρόοδο. Κάναμε μια πρώτη σειρά συζητήσεων με την κυρία Μπαού το Δεκέμβριο για το θέμα αυτό, όταν αντιμετωπίσαμε τα κύρια σημεία που είχαν να κάνουν με τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές προτεραιότητε τη Ουγγρικής Προεδρία. Αλλά βέβαια αυτό ήταν μια συζήτηση σε άτυπο επίπεδο. Και σε ό,τι αφορά τα θέματα της τεχνολογικής πρόοδου, θα πρέπει και στο μέλλον να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα με διτή προσέγγιση και να εγκρίνουμε θέσεις και νομοθετήματα και να ξεκινάμε άτυπες συζητήσεις οι οποίες θα προετοιμάσουν περαιτέρω αποφάσεις γιατί χρειάζονται και για τις έξι που προανέφερα μια κοινή δράση γιατί είναι αλληλέλετες για να μπορέσουμε λοιπόν να καταλήξουμε σε μια κοινή απόφαση για να μπορέσουμε με αποτελεσματικό τρόπο να υλοποιήσουμε όλες τις απαιτούμενες νομικές διαδικασίες μέσα στα, στο εξάμεινο αυτό, θα χρειαστούμε πολλές άτυπες μεταξύ μας συζητήσεις για να μπορέσουμε να προωθήσουμε περισσότερο τα θέματα αυτά. Για το δεύτερο ερώτημά σας, αυτό είναι ένα ε, ερώτημα το οποίο είναι πολιτικό και όχι απλώς οικονομικό, γιατί φυσικά είσαστε και πολιτικοί αλλά και αρμόδιοι για τα θέματα οικονομικής πολιτικής. Και εξάλλου είσαστε και Ευρωπαίοι πολίτες. Για μας είναι απόλυτα σαφές ότι υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης αντιμετώπισης της κρίσης. Δεν υπήρξε αρκετή σύνδεση των δύο διαστάσεων. Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο προφανώς θα πρέπει να ενισχύσουμε και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τους ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς γενικότερα μάλλον, όχι τον ευρωπαϊκό μονάχα και αυτό θα γίνει μονάχα με το να μπορέσουμε να συρρυκνώσουμε τα ελλείμματα του προϋπολογισμού κάτω από το 3%. Η Ουγγαρία μάλιστα έχει δεσμευτεί να το κάνει αυτό. Βάζω και την Ουγγρική μου τραγιάσκα αυτή τη στιγμή για να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε δεσμευτεί να επιτύχουμε ένα έλλειμμα κάτω από το 3% για το 2011. Αλλά αυτή τη στιγμή η περισσότερη προσοχή εστιάζεται στο κρατικό χρέος. Γιατί γενικά σαν μέσος όρο στην ζώνη του ευρώ από 7% πήγε στο 8% και το συνολικό χρέος μπορεί να φτάσει, όχι το έλλειμμα του προπολισμού, αλλά το συνολικό χρέος μπορεί να φτάσει στο 100% του ΑΕΠ. Αν μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυσκολίες, αν μπορέσουμε να θέσουμε τα του οίκου μας σε τάξη και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του κρατικού χρέους στις ε, χώρες μας, νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει μια ευκαιρία να υλοποιήσουμε και να πραγματώσουμε τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Ο Ούγγρος, ως Ευρωπαίος, εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη στρατηγική αυτή η οποία εστιάζει στην απασχόληση, στην παιδεία, στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Και για να κλείσω την απάντησή μου, κυρία Μπάουλ, εμεί ως Ούγγροι είχαμε προτείνει το Συμβούλιο Κοφίν, όταν εγώ ήμουν υπουργό Οικονομικών εκεί, να εστιάσουμε και στην ανάπτυξη και στην απασχόληση και στην, ε, στις ισορροπίες στον προϋπολογισμό, αλλά και την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Το να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, αλλά για να μπορέσουμε να την εξασφαλίσουμε αυτή την ισορροπία, η απάντηση θα πρέπει να εξευρεθεί στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε μια βιώσιμη πολιτική σε σχέση με, την, ε, τα δημοσιονομικά μα με βιώσιμο χρέο και εν καιρό τη μείωση του χρέου αυτού. Τώρα θα πάρουμε τρεις ερωτήσεις. Ούντο πρώτα. Κύριε αναφέρατε τα χρέη των κρατών. Εάν δει κανεί την δομή των χρεών στην Ευρώπη, αντιλαμβάνεται πως δημιουργήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση των δημοσίων προϋπολογισμών λόγω εγγυήσεων χρεοκοπημένων τραπεζών και κερδοσκοπικών Οργανισμό, και εσείς στην Ουγγαρία δείξατε πως είστε σε θέση να βάλετε νέους φόρους όταν η κατάσταση είναι κρίσιμη για να βγείτε από την κρίση. Πότε θα φτάσει η στιγμή να βάλει νέους φόρους στον χρηματοπιστωτικό τομέα η Ευρώπη για να συμμετάσχει και αυτός το τομέα στην αντιμετώπιση της κρίσης. Και δεν θέλετε να ξεκολλήσετε αυτό το θέμα που έχει κολλήσει. Οι Γάλλοι, οι Βέλγοι ήταν υπέρ, η προκατοχή σας, η γαλλική κυβέρνηση είναι υπέρ. Γιατί να φορολογηθούν εκείνες οι τράπεζες οι οποίες έχουν ακόμα ή πολλά υποκαταστήματα, πελάτες ε, και βοηθούν τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά όχι εκείνες οι οποίες κάνουν το λεγόμενο high frequency trading, το οποίο δεν δημιουργεί κάποια αξία, αλλά είναι μόνο κερδοσκοπία και νομίζω πως με ένα πολύ μικρό φόρο μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση στην Ευρώπη. Αν φύγετε, αν σταματήσετε να πατάτε το φρένο, νομίζω θα βοηθήσετε πάρα πολύ εδώ πέρα την κατάσταση. Oui, monsieur le Président. Ευχαριστώ. Το θέμα των ισοτιμιών είναι στο κέντρο της διάσκεψης των J20 που ξεκινάει τώρα. Είπε ότι αποδίδεται μείζωνα σημασία στο μέλλον της Ευρωζώνης, ακόμα κι αν η Ευρωζώνη προς το παρόν δεν είναι μέσα. Η συνθήκη της Λισαβόνας όμως λέει ότι το Συμβούλιο θα ορίζει την πολιτική ισοτιμιών της Ένωσης και όχι η Κεντρική Τράπεζα, ακόμα κι αν η Κεντρική Τράπεζα έχει τα εργαλεία στα χέρια της. Πρώτη μου ερώτηση λοιπόν. Ω εκπρόσωπο του Συμβουλίου θα ζητήσετε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να παρέμβει στην ισοτιμία του ευρώ που κατά τη γνώμη πολλών παρατηρητών είναι υπερτιμημένο σε σχέση με το δολάριο και το γουέν. Αυτό δεν βολεύει και τις εξαγωγές μας αλλά και την ευρωπαϊκή βιομηχανία που υφίσταται τον ανταγωνισμό παραγωγών που βρίσκονται σε χώρες χαμηλού κόστους και όπου το νόμισμα έχει ευθυγραμμιστεί με ένα στενές δολάριο. Δεύτερη ερώτηση. Το ευρωομόλογο. Μας είπατε την ημερήσια διάταξή σας με πολλά θέματα. Δεν είπατε όμως τίποτα για τη συζήτηση για το ευρωομόλογο. Πολλοί θεωρούν ότι το ευρωομόλογο θα ήταν ένα σημαντικό εργαλείο κατά της κερδοσκοπίας παράλογη κερδοσκοπία των αγορών κατά του κρατικού χρέους. Ποια είναι η θέση σας και συμφωνείτε με τον πρόεδρο του Eurogroup σχετικά. Astrid Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν, συγγνώμη και για εσά και για τον Υπουργό για την καθυστέρησή μου. Φταίνουν ε, οι βελγικοί σιδηρόδρομοι. Εγώ είμαι πιστός πελάτης τους, αλλά αυτοί φταίνουν. Κύριε Υπουργέ, με το που έμπαινα στην αίθουσα μιλούσατε για το πρόγραμμα εργασίας σας, το πολύ φιλόδοξο για το εξάμεινο, για το θέμα της ε, φορολογίας των καταθέσεων. Είπατε θέλετε συμφωνία, εκεί που άλλοι μέχρι στιγμής έχουν αποτύχει. Επειδή εγώ είμαι επίκος ενός κράτους που έχει αντιρρήσεις αρχής σχετικά με τις προτάσεις που έχουν γίνει, σας θυμίζω ότι το Λουξεμβούργο δεν λέει πάντα όχι προς όλες τις κατευθύνσεις. Το αποδεικνύει αυτά τα γεγονότα. Είχαμε μια συμφωνία με 27 να συμμορφωθούμε με τα διεθνή πρότυπα σε θέματα πληροφόρησης, δηλαδή ανταλλαγή πληροφοριών, τη αιτήση. Αυτά τα εργαλεία ήδη υπάρχουν και εφαρμόζονται σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς ως Λουξεμβούργοι παίξαμε πλήρως το ρόλο μας στο παιχνίδι αυτό. Το Λουξεμβούργο επίσης συμφώνησε με το Συμβασμό για την διοικητική φορολογική συνεργασία. Όχι δηλαδή ανταλλαγή απόψεων 100% όπως θέλουν μερικοί, αλλά η, η διανοητική τιμιότητα μας επιβάλλει ε, να πούμε ότι ορισμένοι δεν έχουν άρει εντελώ τι αντιρρήσει του. Τώρα, σχετικά με τι διαπραγματεύσει με τι τρίτε χώρε, είναι όρο η Ένωση να φροντίσει να μην βρεθεί υποπινή σε σχέση με τους γειτόνους της. Πρέπει να έχουμε ίδιους κανόνες παιχνιδιού για όλους. Διαφορετικά ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ σε βάρος μας. Επίσης διαπιστώνω ότι αυτές οι τρίτες χώρες και αυτές αλλάζουν τη θέση τους όπως θα ήθελε κατά κάποιο τρόπο η Ένωση Βέβαια τα πράγματα γίνονται βαθμία, αργά-αργά. Αργά αλλά σταθερά. Παραδείγματο χάρη, η Ελβετία, η μεγάλη Ελβετική Συνομοσπονδία, έχει δεσμευτεί σε διμερείς διαπραγματεύσεις με τη Γερμανία και, την, και το Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα φορολογίας καταθέσεων. Και φαίνεται ότι η Ελβετία είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις, σημαντικές μάλιστα. Ας περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα βγει από τις διαπραγματεύσει αυτές, στις λεπτομέρειες τους. Ενδεχομένως μετά και άλλες χώρες μπορεί να τις υιοθετήσουν. Τέλος, κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σα θυμίσω και κάτι άλλο. Το σύστημα που λειτουργήσε πραγματικά και καλά είναι το σύστημα της παρακράτησης στην πηγή. Ανταλλαγή πληροφοριών. Το θέμα είναι κάπως φλού. Δεν ξέρουμε αν πραγματικά έχει σημειωθεί πρόοδος de facto. Αυτό ήθελα να σας πω κύριε Υπουργέ και ελπίζω στην Προεδρία σας να στεφτείτε με επιτυχία, από επιτυχία. Και να λάβετε υπόψη τα σχόλιά μου. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε τον κύριο Υπουργό να απαντήσει. Ευχαριστώ. Κύριε Μπούρμαν. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη δερμηνία. δεν ακούγεται η δερμηνία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 Ίσως να είναι συμβολικό αυτό που συνέβη. Όταν μιλάμε δηλαδή για τον φόρο προς τις τράπεζες, η τεχνολογία δεν ακολουθεί. Η Ουγγαρία και, πρώτη και μετά ε, το Ηνωμένο Βασίλειο εισήγαγε αυτόν τον φόρο των τραπεζών από πέρυσι. Μεγάλες συζητήσεις, μεγάλες αντιρρήσεις Τώρα 10 περίπου μέλη της Ένωσης έχουν ένα είδος, κάποιο είδος φορολόγηση των τραπεζών. Υπάρχουν μεταβατικές διατάξεις, υπάρχουν όμως και φόροι οι οποίοι έχουν μπει στο δρόμο τους με μακρόπνοη προοπτική σε μερικά κράτη-μέλη. Η εισαγωγή του τραπεζικού αυτού φόρου είναι επικίνδυνη, μια επικίνδυνη απόφαση. μπορεί οι τράπεζε, παραδείγματο χάρη, να σταματήσουν να κάνουν επενδύσει. Βέβαια, όλε οι 10 χώρε μέλη που ανάφερα που είπα ότι εφαρμόζουν τέτοιου είδου μέτρα παρουσίασαν επιχειρήματα, μερικά πάρα πολύ σοβαρά επιχειρήματα οικονομικής πολιτικής, με βάση τα οποία προκειμένου να πετύχουμε οικονομική ανάπτυξη, να έχουμε νέα απασχόληση, νέες επενδύσεις κεφαλαίου, καταρχήν θα πρέπει να μπει τάξη στον προπολογισμό, να σταματήσει η τάση αύξησης του εθνικού χρέους και των εθνικών ελλημάτων. Για να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης που είχε η Ένωση μέχρι και πρόσφατα, πρώτα πρέπει να μπει τάξη στα δημόσια οικονομικά, στον προπολογισμό, να σταματήσει να αυξάνεται το χρέος και από τη στιγμή που θα το έχει πετύχει αυτό μια χώρα, τότε μπορεί να κοιτάξει τα της ανάκαμψης. Βέβαια, αυτά τα επιχειρήματα είναι σεβαστά. Και νομίζω σε όλες τις χώρες μέλη, όπου εφαρμόζεται φορολόγηση των τραπεζών, από όσο ξέρω τουλάχιστον εγώ, σε όλες τις χώρες αυτές αυτός ο φόρος συνοδεύεται και από άλλα μέτρα οικονομικής πολιτικής με συγκεκριμένους στόχους. Υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά τις επενδύσεις και τη δημιουργία απασχόλησης. Αυτά τα δύο κινούνται παράλληλα. Διαφορετικά ε, θα υπερισχύσει μόνο ο κίνδυνος λόγω της φορολόγησης των τραπεζών. Η σύσταση της Προεδρίας μας είναι να επεξεργαστούμε ένα σύστημα φορολόγησης των τραπεζών με διάφορες παραμέτρους, εναρμονισμένο ή δυνατόν σε κοινοτικό επίπεδο. Προχωρώ στο επόμενο μιλητή που, που έθεσε δύο ερωτήσεις. Ως οικονομολόγος, ούτε στην Ουγγαρία, ούτε στο ΕΚΟΦΗΝ, δεν θα όριζα στόχους ισοτιμιών. Αυτό πρέπει να καθορίζεται από τις χρηματαγορές και από τις ανεξάρτητες τράπεζες, τις εκδότριες τράπεζες, τις κεντρικές. Αυτό είναι θέμα Αυτό αφορά και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία είναι ανεξάρτητη Ο πρόεδρος του ΕΚΟΦΗΝ και άλλοι πολιτικοί δεν θα έπρεπε να διαμορφώνουν γνώμη ή συστάσεις σχετικά με οτιδήποτε αφορά την ισοτιμία. Η δουλειά μας είναι να δημιουργήσουμε ένα σωστό περιβάλλον οικονομικής πολιτικής όπου άσχετα με το ποια είναι η ισοτιμία να οδηγούμαστε σε οικονομική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων Διότι αν δεν συμβεί αυτό, αν δεν έχουμε οικονομική ανάπτυξη, αν δεν έχουμε απασχόληση, αν δεν έχουμε δημογραφική ανάπτυξη, παιδιά και ε, επενδύσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλα τα άλλα δεν φτουράνε. Δεύτερη ερώτησή σας, ευρωομόλογα. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλή ιδέα. Αλλά πριν το εκδώσουμε, το ευρωομόλογο στην Ευρωζώνη, ή προαπειλεί δημιουργίσμο μιας γωαράς ευρωμολόγων. Θα πάμε βάλουμε ταξί στα σπίτια μας. Αυτό είναι προτεριότητα της Ουγρικής προεδρίας και ήπαυρην η πριν δημιουργήσουμε μια αγορά ευρωμολόγων, θα πρέπει να βάλουμε τάξη στα σπίτια μας. Αυτό είναι προτεραιότητα της Ουγγρικής Προεδρίας. Και είπα πριν, η οικονομική διακυβέρνηση, αλλαγή των συνθηκών, ευρωπαϊκό εξάμεινο, ο μηχανισμός σταθεροποίησης. Όλα αυτά τα εργαλεία είναι αναγκαία για να ενισχυθεί το ευρώ η Ευρωζώνη και η Ένωση τελικά. Από τη στιγμή που θα το έχουμε πετύχει αυτό, ως ισχυροί παίχτες θα είμαστε σε θέση να φτιάξουμε και μια αγορά ευρωμολόγων. Και για να έχουμε τέτοια αγορά χρειαζόμαστε μια στιβαρή οικονομία, φερέγγια. Ευχαριστώ για τα ευγενικά λόγια της κυρίας Λουλή. Η Ουγγρική Προεδρία στο ΕΚΟΦΗΝ θα συμβάγει σε λύση. προκειμένου να αρθούν ακόμα τα εκκρεμή θέματα της ε, οδηγίας για τη φορολόγηση των καταθέσεων έχουμε ορίσει στόχο μας πολιτική συμφωνία. Φαίνεται να υπάρχουν δύο θέματα εκκρεμή και τα δύο είναι πολιτικής φύσης. Το ένα είναι οι εξωτερικές συνθήκες, οι εξωτερικοί όροι και το άλλο είναι η μεταβατική φάση. Προσωπικά και το κάναμε ήδη, κινήσαμε μια διαδικασία διμερών συζητήσεων με τις ε, χώρες μέλη και τους αντίστοιχους υπουργούς τον οποίο χρειαζόμαστε τη βοήθεια προκειμένου να πετύχουμε μια κοινή πολιτική συμφωνία. Η Αυστρία, το Λουξεμβούργο και η Δανία, η Ιταλία, η Γαλλία και φυσικά το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σουηδία θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν όλοι αυτοί οι υπουργοί να συμφωνήσουν και από τη στιγμή που θα το έχουμε πετύχει αυτό και αυτό θα προσπαθήσουμε εμείς να πετύχουμε με τις διμερείς συζητήσει, τότε ίσως μπορέσουμε να πετύχουμε την πολιτική συμφωνία για την οδηγία αυτή φορολόγησης των καταθέσεων. Αυτά αυτό είναι μια από τις σημαντικές πρωτοβουλίες της Προεδρίας μας. Τέσσερις ακόμα έχουν <clears throat> μείνει που θέλουν να θέσουν ερωτήματα. Ε, η Σίλβη και ο Φιλίπ. Στο τέλος, στο τέλος ούτω. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Κάτι πάρα πολύ απλό θέλω να σας ρωτήσω. Εδώ είμαι. Ως μία από τις εισηγήτριες για αυτή τη δέσμη μέτρων, σας πενθυμίζω ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του πρόσφατα είπε ότι είναι απαραίτητο να επιταχυνθούν οι εργασίες για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλω να φέρω την προσοχή σας στο γεγονός ότι μπορούμε να κινηθούμε ταχύτερα και να έχετε μεγαλύτερη επιτυχία και σαν Ουγγρική Προεδρία, αν μπορέσει να υπάρχει μια παγιοποίηση της θέσης του Συμβουλίου ανεξάρτητα από αυτά τα οποία πράττει το Κοινοβούλιο, το οποίο φυσικά θα πρέπει να λάβει υπόψη και τη θέση του Συμβουλίου. Θέλω να πιστήσω λοιπόν την προσοχή σας στο ότι στις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αποφύγετε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να κινηθούν σε αντίμαχες κατευθύνσεις, γιατί αλλιώς ο χρονικός ορίζοντας του Ιουνίου δεν θα είναι επαρκής. Το θέμα των ευρωμολόγων το ανέφερα και στην εκθεσή μου, γιατί νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιληφθούμε αυτού του θέματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή μας και φυσικά και στην Ολομέλειά μας. Είπατε ότι είναι απαραίτητο να τακτοποιήσει ο καθένας τα του οίκου του, φυσικά. Αλλά, και αυτό είναι το πνεύμα των προτάσεών μου, δεν θα πρέπει να υπάρχει σύγκρουση μεταξύ μιας πειθαρχία και μιας αγοράς <clears throat> ρευστής σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πειθαρχία λοιπόν και η δημιουργία προσφόρων εργαλείων δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έρθει σε σύγκρουση θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η άποψή για αυτά που είπε ο Τσέκερ και ο Μπρούγκελ για, τους μπλε και κο... για τα μπλε και τα κόκκινα ομόλογα όπω αναφέρονται. Αν θεωρείτε λοιπόν ότι αυτά τα εργαλεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να υπάρχει μια μεγαλύτερη τάση συμμόρφωση προ του κανόνε. Αντίθετα με αυτά που είχα πει ο κύριος Λάγκεν και ο κύριος Κάρης είπανε τελευταία στιγμή ότι θέλουν να λάβουν το λόγο ο Φιλίπ και μετά η Κορίν. Σας ευχαριστώ λέει ο Φιλίπ. Εδώ είμαι. Θέλω να αντιμετωπίσω καταρχήν το θέμα της φορολογίας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι απαραίτητο να επιτύχουμε και κάποια σύγκληση στον τομέα της ε, φορολογίας αν θέλουμε να έχουμε μια κάποια συνεκτικότητα και να συνεχίσουμε να έχουμε τη δυνατότητα επενδύσεων. <clears throat> Υπήρξε μια πρόταση που αναφέρθηκε ήδη από τον Ούντο για το πώς να φορολογηθεί ο χρηματοοικονομικός τομέας. Υπάρχει η πρόταση γνωστή αυτή για το φόρο χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Και μετά υπάρχει πάλι μια άλλη έννοια, μια άλλη σύλληψη που έχει να κάνει με τον φόρο χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Δεν ξέρω ποια είναι θέση για το θέμα αυτό, θα ήθελα να το ξέρω. Δεύτερον, η Ουγγαρία, και μερικές φορές μπορώ να είμαι και θετικός μαζί σας, έχετε αναλάβει την ε, θαραλέα αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση της φορολογίας των ε, πολυεθνικών επιχειρήσεων. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχει σωστή φορολογία των πολυεθνικών οργανισμών σε όλη την Ευρώπη και φυσικά υπάρχει το θέμα της ενεργειακής φορολογίας και της αντιμετώπισης φοροδιαφυγής. Το ερώτημα μου είναι απλό, αλλά νομίζω ότι είναι απλό και να το απαντήσετε. Ποια είναι, ποια είναι η πρακτική και συγκεκριμένη στόχη που θα σας επέτρεπαν εσείς να θεωρήσετε ότι η Ογγρική Προεδρία έχει επιτύχει σε σχέση και με τους τέσσερις στόχους και πώς θα τους αντιμετωπίσετε τους στόχους αυτούς, ποια είναι η στρατηγική σας. Επίσης αναφερθήκατε πολλές φορές στο κρατικό χρέος, <clears throat> αλλά και το ιδιωτικό χρέος πολλές φορές είναι ένα ακόμα πιο σημαντικό θέμα. Σημερίζεστε μια τέτοια άποψη και εάν ναι, τι θα μπορούσε να γίνει για το ιδιωτικό χρέος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης θα ήθελα να συνεχίσω αυτά που είπε η Σιλβή. Ναι, να βάλουμε τον Νίκο μας σε τάξη, αλλά μετά να δούμε πώς και πού θα επενδύσουμε. Είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να το κάνουμε αυτό μαζί, γιατί ο κόσμος δεν θα περιμένει να τακτοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κόσμος συνεχίζει να κινείται. Και εμείς χάνουμε συνέχεια ανταγωνιστικότητα και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Πρέπει να επενδύσουμε και να συνεχίσουμε να επενδύουμε, ενώ συνεχίζει αυτή η διαδικασία τακτοποίησης των εσωτερικών της Ευρώπης. Η Κορίνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αφαιρθώ σε αυτό το οποίο είπε η Σιλβί Γκουλάρ για την διαδικασία για το πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Είναι κρίσιμη σημασία στο Συμβούλιο να ακούσει την άποψη του Κοινοβουλίου όσο το δυνατόν νωρίτερα, γιατί αν θέλετε να έχουμε συμφωνία τον Ιόνιο, πρέπει να γίνει αυτό εξ αρχής. Και θα ήθελα άρα να υπογραμμίσω αυτό το οποίο είπε η Σιλβί, για το πως δεν θα πρέπει να είναι πολύ άκαμπτη η θέση του ΕΚΟΦΗΝ πριν γίνει ο διάλογος με το Κοινοβούλιο. Για το Κοινοβούλιο έχει ουσιαστική σημασία πρώτα απ' όλα να έχουμε εντολή από την Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων για να συνομιλήσουμε με την Προεδρία και ελπίζω να το αντιληφθείτε αυτό και βέβαια θα μπορούσαμε να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι εάν είχε εμπλακεί στη διαδικασία της Task Force στο Κοινοβούλιο. Οπότε ελπίζω πως θα σεβαστείτε το Κοινοβούλιο και τη θέση του Κοινοβουλίου εδώ πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επαναλάβω πως ο κύριος Μπούλμαν ρώτησε συγκεκριμένα το εάν η Ουγγρική Προεδρία θα υποστηρίξει τον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών όπως έκανε και η Βελγική Προεδρία. Φαντάζομαι πως εδώ παραθέλει ένα ναι ή ένα όχι. Και ο Φιλίπ το ίδιο ρώτησε. Οπότε αν θέλετε να απαντήσετε σε αυτή τη σειρά ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Να απαντήσω καταρχήν στην κυρία Γκούλαρτ. Όταν μιλάμε για επιτάχυνση των εργασιών σχετικά με τις έξι νομοθετικές προτάσεις όπου απαιτείται κοινή απόφαση εννοούμε ότι όλες οι τυπικές και άτυπες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πλήρως, που σημαίνει χρειάζονται έξυπνοι συμβασμοί, όλοι τους χρειαζόμαστε. Αυτή η δουλειά πρέπει να επιτεχυνθεί. Δεν είναι μια διαδικασία που πρέπει να γίνει στο πόδι. Χρειαζόμαστε έξυπνους συμβασμούς, όπως είπα, που σημαίνει καλά προετοιμασμένες αποφάσεις, και τυπικά και άτυπα και συμφωνώ με την κυρία Γκουλάρ ότι είναι της αρμοδιότητας των εθνικών κυβερνήσεων και διάφορα μέτρα που, έχει πάρει, που έχουν λυθεί στην Ευρωζώνη όλα αυτά πρέπει να κινηθούν παράγγελα. Όσον αφορά τον φόρο στις τράπεζες, επιτρέψτε μου να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα, αναφέροντας τον Keynes. Σε χαλιπούς καιρούς, όπου χρειάζεται ο φόρος στις τράπεζες και 10 χώρες έκριναν ότι χρειάζεται αυτός ο φόρος, σε χαλεπούς καιρούς λοιπόν λέω, αυτό θα είναι για να μπει σε τάξη το δημοσιονομικό έλλειμμα. Αυτό σημαίνει ότι στους καιρούς που ζούμε, ο φόρος αυτός θα πρέπει να υποστηρίξει την εξυγίανση των κρατικών προϋπολογισμών. Στους καλούς καιρούς των παχιών αγελάδων, ο φόρος στις τράπεζες θα είναι για να δημιουργήσει ένα αποθεματικό για τους επόμενους καλεπούς καιρούς. Σας θυμίζω ότι ο John Maynard Keynes είπε ότι στους κακούς καιρούς πρέπει να, να δαπανούμε περισσότερα όσο γίνεται και τους καλούς καιρούς, τον καλό καιρό να βάζουμε κάμποσα χρήματα στην άκρη για τον κακό καιρό. Στη δεκαετία του 90 και μετά, στην αρχή, πιστεύαμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία κρίση οικονομική, χρηματοπιστωτική κλπ. Όπως λέγανε οι Αμερικάνοι ότι θα υπάρξει. Στις 7 Απριλίου είχαμε τις πρώτες γνωστές καταρρεύσεις και μεταξύ του 2001 και 2003 είδαμε την Αμερικάνικη κρίση. Τον Οκτώβριο είδαμε να εμφανίζεται μια άλλη είδους κρίση να αφορά λοιπόν τον φόρο στις τράπεζες, εγώ προτείνω να έχουμε κατά νου αυτά που είπε ο Κέινς. Δηλαδή να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά μας, τον προπολογισμό μας και στο μεταξύ να το χρησιμοποιήσουμε για να βοηθηθούμε να ξεπεράσουμε την κρίση, να μην χαθούν και άλλες θέσεις απασχόλησης να χρησιμοποιηθεί λοιπόν αυτός ο φόρος. Όταν όμως θα αρχίσει πάλι να λάμπει ο ήλιος, να το χρησιμοποιούμε ως εργαλείο αποτροπής της επόμενης κρίσης. Και αν αυτό συμβεί, ας ελπίσουμε ότι δεν θα συμβεί και ότι δεν θα είναι τόσο καταστροφική όσο η κρίση που ζούμε σήμερα, να έχουμε ένα καλό απόθεμα να βοηθηθούμε στην νέα αυτή κρίση. Ευχαριστώ πολύ για το ότι αναφέρατε την περικοπή του φόρου ε, στις επιχειρήσεις στην Ουγγαρία. Το κάναμε αυτό για να υποστηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την 1η Ιουλίου εισήχθη αυτός ο νόμος. Οι πρώτες αντιδράσεις ήταν θετικές και πιστεύουμε ότι πρέπει να περικόψουμε και τον φόρο εισοδήματος και να αυξήσουμε άλλου είδους πηγές εισοδήματος για να δημιουργηθεί επιπλέον απασχόληση και επενδύσεις. Βέβαια, σχετικά με τις επενδύσεις των πολιεθνικών, η Ένωση έχει νομοθεσία, έχει κανονισμό, ο οποίος πρέπει να τηρείται από όλους. Συμφωνώ ότι ο κόσμος δεν πρόκειται να μας περιμένει. Να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε τους προπολογισμού και το χρέος. Στο μεταξύ χρειαζόμαστε οικονομική ανάπτυξη, επενδύσεις, απασχόληση. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας ταυτόχρονα και πιστεύω ότι το Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ επικεντρώνεται κυρίως σε εργαλεία δημοσιονομικής εξισορρόπησης. Οικονομική διακυβέρνηση, πρόληψη και ε, διορθωτικά μέτρα. Τα άλλα συμβούλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως Συμβούλιο Ανταγωνισμού Φερπίν, εκεί προγραμματίζεται το θέμα των επενδύσεων, ας πούμε, για την επόμενη δεκαετία. Επίσης συμφωνώ με το ότι το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο αλληλοεξαρτώνται. Επαναλαμβάνω κάτι που είπα και πριν. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλους, όλες τις μεθόδους, τυπικές και άτυπες, να φτιάξουμε γέφυρες ανάμεσα στα τρία όργανα. Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο. Και να δημιουργήσουμε την οικονομική δομή των έξι νομοθετικών προτάσεων έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν από το τέλος Ιουνίου και μετά. Για τον κύριο Μπούλμαν, ο οποίος έκανε μια δεύτερη ερώτηση, μια επιπλέον ερώτηση ποια είναι η γνώμη μου για τον επικεφαλής ε, του Συμβουλίου ΕΚΟΦΗΝ για τον φόρο στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε μια πολύ εμπεριστατωμένη ανάλυση και μετά να αποφασίσουμε για το χρηματοπιστωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένου και των χρηματιστηρίων, τον ασφαλιστικό κλάδο, μόνο μετά να πάρουμε, αν πάρουμε απόφαση για νέους φόρους. Γιατί όσον αφορά τον φόρο επί των συναλλαγών, η Ένωση είναι ένας μόνο από τους παίκτες. Είναι βέβαια από τους μεγάλους παίκτες στην παγκόσμια οικονομία, αλλά αν θέλουμε να πετύχουμε μια κοινή συμφωνία στο επίπεδο των G20, σχετικά με τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, αυτό θα δημιουργούσε ασφάλεια για όλη την Ένωση. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε υπόψη κατά νου δύο τινά. Πρώτον, η κρίση προήλθε από το χρηματοπιστωτικό κλάδο. Το δεύτερο, πρέπει να εισαχθεί νέα φορολογία μόνο αν αυτή η νέα φορολογία μας εξυπηρετεί. Και γι' αυτό πρέπει να γίνει πρώτα μια εμπεριστατωμένη ανάλυση πριν εισαχθεί, πριν επιβληθεί ένας τέτοιου είδους φόρος. Αυτό αφορά και τον φορολόγηση των τραπεζών και τον φόρο στις συναλλαγές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω πως Βεβαίω, το ζήτημα τη ταχύτητα έχει προκύψει σε πολλέ ε, ιδιωτικέ συναντήσει που είχα. Καθώ λοιπόν μεταδίδεται η συνεδρία στο διαδίκτυο, θα επαναλάβω αυτό το οποίο έχω πει πολλέ φορέ, πω εμεί, ε, η Επιτροπή μα έχει μόνο μία ταχύτητα, η οποία είναι γρήγορη και συχνά παραπονιούνται οι άλλε επιτροπέ. Οπότε δεν σκοπεύουμε να χασομερίσουμε και θα κάνουμε τη δουλειά μας επιμελώς αλλά με τη συνήθη ταχύτητα. Τέσσερις λοιπόν ομιλητές ε, ε, έχουν απομείνει στη λίστα γιατί συνεχώς μεγαλώνει. Οπότε Βέρνε Λάγγεν, Οτ Μαρκάρας, ο κύριος Τούσας και Πέρες. Θα σας ακούσουμε όλους λοιπόν. Βέρνερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Έχω ένα ερώτημα για τις διαβουλεύσεις στην ομάδα εργασίας Συμβουλίου. Εδώ, εδώ πέρα κάθομαι στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου με θέμα ρύθμιση των παραγόγων. Μετά την πρόταση της Βελγικής Προεδρίας που ε, έκανε δεκτή και η Ουγγρική, βλέπουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο, από ό,τι φαίνεται, δεν θα συμπεριλάβει μόνο τα παράγωγα εκτός χρηματιστηρίου αλλά όλα τα παράγωγα στο πεδίο εφαρμογή Μέχρι στιγμής δεν είχαμε δημόσια συζήτηση ούτε αιτιολόγηση για αυτή την κίνηση. Δεύτερον, σε αντίθεση με αυτό, ε, βλέπουμε πως ζητούνται όλο και περισσότερες εξαιρέσεις. Είτε μιλάμε για εμπόριο ενέργειας, ε, ταμεία συντάξεων, ε, δημόσιες τράπεζες, τομέα ακινήτων. Όλοι θέλουν από μία εξαίρεση. Και τρίτον, Θεωρώ πως ε, το μητρό αυτό συναλλαγών ε, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν έχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και για τα παράγωγα. Μόνο έτσι μπορεί να συμπεριληφθεί και αυτό το μέτρο για τις ιδιωτικές ε, συναλλαγές και υπό κάποιες συνθήκες να δημοσιευτεί. Τώρα ακούμε από το Συμβούλιο πως υπάρχει ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για να υπάρξει μια κοινή θέση σε ένα δύσκολο θέμα που περιλαμβάνει ακόμα 11 ζητήματα επίμαχα και αυτό θέλετε να το έχετε ολοκληρώσει μέχρι το Συμβούλιο του Μαρτίου την Ιαρινή Σύνοδο. Θέλετε να μας πείτε πώς θα το κάνετε αυτό και ταυτόχρονα να λάβετε υπόψη και τη θέση του Κοινοβουλίου. Γιατί βρισκόμαστε στη διαδικασία της συναπόφασης και Βεβαίως ε, εμείς ε, στηρίζουμε σε μεγάλο βαθμό την θέση της Κομισιόν και αν πάει σε άλλη κατεύθυνση το Συμβούλιο θα έχουμε σοβαρή αντιπαράθεση ε, που δεν νομίζω να μπορέσει δηλαδή να λυθεί επί Ουγγρικής Προεδρίας. Ναι, κύριε Υπουργέ, έχω την εξερώτηση σύντομα. Πρώτο θέμα, θα ήθελα να μάθω από σας πότε οι Υπουργοί Οικονομικών θα σταματήσουν το μπλοκάρισμα της Κομισιόν για την ομπρέλα αυτή προστασίας και πότε μπορούμε να υπολογίζουμε σε εμβάθυνση και διεύρυνση αυτής της ομπρέλας προστασίας. Τρίτον, πήγαμε από ένα διακυβερνητικό σε ένα κοινοτικό όργανο με εμπλοκή Κοινοβουλίου Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δικαστηρίου όσον αφορά αυτή την ομπρέλα προστασία. Κατόπιν μιλήσατε για φόρο στις τράπεζες. Μήπως ε, ακριβώς το παράδειγμα της Ουγγαρίας μας δείχνει πως οι διαφορετικές ε, φορολογίες των τραπεζών οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού και θα έπρεπε να έχουμε μία ενιαία φορολογία. Και είχατε εσείς αυτό το ειδικό τέλος των ε, τραπεζών το οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί αντίθετο προς το ευρωπαϊκό δίκαιο εάν αφορά μόνο τις ξένες τράπεζες και όχι τις ε, εγχώριες. Ευχαριστώ. Κύριος Τούσας μετά. Για το 2010 το ακαθάριστο δημόσιο χρέο τη ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε συνολικά στο 85% περίπου του ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ και σε 80% σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αποτέλεσμα να προσθεθεί η δημοσιονομική επιβάρηση 4,5% στο ΑΕΠ μακροπρόθεσμα. Συνολικά το 9,6% του ενεργού πληθυσμού είναι άνεργοι. Σε ορισμένες χώρες η ανεργία των νέων φτάνει στο 40%. Περίπου 80 εκατομμύρια άτομα υπολογίζεται ότι διαβιούν κάτω του ορίου φτώχεια στην Ευρώπη. Θα ήθελα με την ευκαιρία τη σημερινή σα παρουσία στην Επιτροπή να ρωτήσω το εξή. Μπορείτε να μα ενημερώσετε αν στα πλαίσια τη Ουγγρική προεδρία ή στο ΕΚΟΦΗΝ συζητούνται τα εξής θέματα. Σε ό,τι αφορά τις χώρες που έχουν μεγάλο χρέος. Πρώτο, επιμήκυση του χρόνου εξόφλησης του χρέους. Δεύτερο, μείωση των επιτοκίων δανεισμού. Και τρίτο, αναχρηματοδότηση του χρέους από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό. Ευχαριστώ. Okay. Very quickly, Vicky, and then uh, yes, just coming back on what you... Ναι, για να επανέλθω σε αυτό το οποίο είπατε για τους φόρους επί των τραπεζών και αναφέρατε τον Κέινς βεβαίω, ο οποίος είχε εξηγήσει πως σε δύσκολους καιρούς πρέπει να εξοδεύουμε περισσότερο. Όπως αντιλαμβάνομαι εγώ βεβαίως, τον Κέινς είναι πως θα πρέπει να εξοδεύουμε. Ε, σε κακούς καιρούς γιατί δεν μειώνονται οι μισθοί. Αλλά βλέπουμε σε αυτή την ε, κρίση στον ιδιωτικό τομέα πώς μειώνονται οι μισθοί. Δεν έχουμε δει το ίδιο πράγμα στο δημόσιο τομέα. Ποια είναι η άποψή σας λοιπόν για τις ε, αυξανόμενες αποκλήσεις όσον αφορά τις προσδοκίες εργαζομένων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ και για τις απαντήσεις που δώσατε και τα σχόλιά σας. Όλοι γνωρίζουμε και εσείς ξέρετε πως δεν μπορεί να γίνει κανένα θαύμα μέσα σε έξι μήνες, αλλά πρέπει να ορίσουμε σωστές προτεραιότητες. Είναι προς ε, το συμφέρον μας αυτό. Και έτσι θα διασφαλίσουμε πως ε, θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Πράγματι δεν υπάρχει κανένα απλός τρόπος, δεν υπάρχει κανένα θαύμα που μπορεί να γίνει ούτε για τον φόρο χρηματοοικονομικές συναλλαγής, ούτε για το ευρωομόλογο. Όμως Εγώ είμαι ευγνώμων για το ότι η Ουγγρική Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ε, γνώμη των μέλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τέσσερα πράγματα αναφέρθηκαν ως βασικά σε σχέση με την οικονομική πολιτική, όμως η έμφαση που δίδεται δεν είναι η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη, οπότε δεν υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Μιλήσατε για την ισορροπία, την ε, ανάπτυξη και την απασχόληση και το δημογραφικό ζήτημα. Βεβαίω ε, όλα αυτά δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ε, ταυτόχρονα. Είχατε ένα καλό σχέδιο το οποίο ήταν το σχέδιο Σίτζενη μεταξύ 1998 και 2000 οδήγησε σε ανάπτυξη. Πώς θα μπορεί να μας βοηθήσει λοιπόν κάτι τέτοιο σε έναν κλάδο που είναι ίσως ο κινητήρας της οικονομίας και της απασχόλησης και αναφέρομαι βεβαίως εδώ πέρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι η εγγύηση για το μόνο. και πώς θα συσχετιστεί αυτό με το σχέδιο για την Ευρώπη 2020. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση που έγινε για τα παράγωγα. Ξέρετε πως ε, τα παράγωγα over the counter σκοπεύουμε πρώτα απ' όλα εκεί πέρα να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Οπότε, χωρίς ε, διαφάνεια, ξέρετε πως ε, μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα στο, στο ημίφος. Οπότε, στόχος μας είναι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί στο πλαίσιο των G20 από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να πραγματοποιηθούν και βεβαίως μπορούμε να φτιάσουμε σε μια λύση ανάλογη με αυτή που έχει εφαρμοστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγματι λοιπόν χρειάζεται μια γενικότερη προσέγγιση και θέλουμε να ολοκληρωθεί ε, η προσέγγιση μας τον Μάιο, να έχουμε ένα πλαίσιο συμφωνίας. Και ε, για τα παραγωγά over the counter και για αυτά τα οποία διακινούνται μέσω χρηματιστήριου. Μετά, ο κύριος Κάρας. Να... Θα ήθελα, δεν ξέρω αν μπορείτε να αναδιατυπώσετε το ερώτημά σας για την ομπρέλα προστασίας. Αλλά για το θέμα της φορολογίας των τραπεζών να απαντήσω κάπως σύντομα. Κάποιες χώρες βρήκαν κάποιες λύσεις φορολογώντας τις τράπεζες. Βεβαίω, η περίπτωση την οποία γνωρίζω καλύτερα είναι η Ουγγρική. Στην ε, περίπτωση λοιπόν της δικής μας ε, της φορολογίας δεν κάνουμε διάκριση μεταξύ ξένων και χώριων τραπεζών κατά κανέναν τρόπο. Στην ε, Ουγγαρία ο φόρος επί των τραπεζών αφορά οποιαδήποτε εταιρεία δραστηριοποιείται στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείε, εταιρείε ε, χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Και επειδή στην Ουγγαρία η μεγαλύτερη τράπεζα είναι ουγγρική ιδιοκτησία, αυτή πληρώνει και το περισσότερο φόρο. Έτσι είναι τα πράγματα, απλώς όταν δεν κάνουμε καμία διάκριση με βάση την ιδιοκτησία της τράπεζας. Τώρα, ε, μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημά σας για την ε, ομπρέλα προστασίας. Είναι... Ήθελα να μου πείτε πότε σκοπεύετε να, πότε βλέπετε να λάβετε απόφαση για την πρόταση της Κομισιόν για τη διεύρυνση της ομπρέλας προστασίας. Γιατί αναβλήθηκε την τελευταία Δευτέρα και δεν ξέρω αν θεωρείτε πως θα πρέπει να γίνει κοινοτική και να βγει από εκεί το διακυβερνητικό στοιχείο. Ευχαριστώ. Τώρα, κατάλαβα Λοιπόν, και το Συμβούλιο Εκοφήν ε, και τα άλλα θεσμικά όργανα συνεργάζονται για να δημιουργήσουν ένα μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας, αλλά δεν ε, έχουμε κάποια αρμοδιότητα να λάβουμε απόφαση στο πλαίσιο του ΕΚΟΦΗΝ ούτε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε συμμετέχουμε εμείς, λέμε τις απόψεις μας, αλλά είναι τελείως διακυβερνητικό το ζήτημα. Οπότε ο κύριος Γιούνκερ, ε, εκπροσωπώντας την Ευρωζώνη, έχει την πρωτοβουλία Οπότε στο πλαίσιο του ΕΚΟΒΗΝ, του ΕΚΟΦΗΝ τα βλέπουμε αυτά τα ζητήματα, είναι πολύ σημαντικά. όσον αφορά τις προτεραιότητες μας, αλλά όπως σας είπα είναι κάτι το οποίο θα, θα λυθεί με διακυβερνητική απόφαση. Οπότε Κύριε Τούσα, τώρα η κατάσταση που περιγράφεται είναι πολύ γνωστή σε εμά. Έχουμε ανεργία πάνω από 10%, αυξανόμενο δημόσιο χρέο και ω αποτέλεσμα αυτών μικρή ανάπτυξη. Ε, είναι γνωστό το σενάριο. Ε, ίσως να μην αλλάξει να μην αλλάξει σε ένα εξάμεινο τα πράγματα, αλλά έχουμε το μηχανισμό σταθερότητας και με τις υπόλοιπες προτάσεις καταφέρουμε να γυρίσουμε την κατάσταση. Αυτό το οποίο έχει σημασία κατά την απόψή μου εδώ πέρα είναι το ότι παρά το ότι έχουμε κοινά ή παρόμοια προβλήματα και οι 27 χώρες μέλη και βεβαίως οπωσδήποτε οι χώρες της ε, Ευρωζώνης πάρα πολύ συχνά υπάρχουν ε, Συγκεκριμένε, εξειδικευμένε λύσεις που μπορεί να εφαρμοστούν. Οπότε σε ένα γενικότερο πρόβλημα ε, μπορεί να μην έχουμε μία ενιαία λύση. Οπότε μέχρι το τέλος Μαρτίου πρέπει να καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις οι οποίες θα αφορούν συγκεκριμένα το κάθε κράτο μέλος και εκεί πέρα θα συζητηθούν τα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που θα βοηθήσουν τα κρατημένα να αντιμετωπίσουν το κοινό αυτό πρόβλημα. Πρέπει να παραδεχτώ πως δεν είμαστε βεβαίως μέλο τη Ευρωζώνης αλλά εντός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν είναι να σταθούμε έναντι του ανταγωνισμού από την Ασία και τη Βόρεια Αμερική, τα προβλήματα είναι κοινά. Ξέρετε πως έχουμε ένα ποσοστό απασχόλησης γύρω στο 65%, στη ΣΥΠΑ είναι 75%, ενώ στις χώρες της Ασίας, στην Κίνα, είναι ένα 85% το ποσοστό απασχόλησης. Οπότε στην Ευρώπη πρέπει να, να δούμε αυτό το πρόβλημα. Η χαμηλή ρυθμή ανάπτυξης τα υψηλά χρέη και το χαμηλό ποσοστό απασχόλησης. Το οποίο βεβαίως ε, συμπίπτει και με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Οπότε πρέπει να έχουμε απαντήσεις οι οποίες ε, θα είναι εξειδικευμένες στην κάθε χώρα και θα αφορούν τα προγράμματα δομικών μεταρρυθμίσεων. Για αυτά τα προγράμματα δεν δομικών μεταρρυθμίσεων δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν με μία συνταγή, γιατί είναι πολύπλευρη η Ευρώπη και πολύπλευρη είναι και η απάντηση την οποία χρειαζόμαστε στα προβλήματα αυτά. Όσον αφορά δε τον Κέινς, αγαπητή κυρία, ο ιδιωτικός τομέας αντέδρασε πιο γρήγορα και η αντίδραση του ιδιωτικού τομέα ήταν γύρω στο ήταν μια διαφορά φάση θα έλεγα νέα μηνών. Οπότε όταν έχουμε μια ανάκαμψη και θα αντικατοπτριστεί, αυτή, θα στα νούμερα δεν θα συμπέσει αμέσως ε, με αύξηση της ε, απασχόλησης και οπωσδήποτε όχι στον ε, δημόσιο τομέα που είναι κάπως αργότερος στον να αντιδράσει εξελίξεις. Την τελευταία δεκαετία θα ήμασταν επιτυχείς σε αυτό το οποίο όπως είπε ο Κέιντς. Και βεβαίω θα έπρεπε να είχαμε κάνει αυτό το οποίο έλεγε πω ε, στου καιρού των παχαίων αγελάδων καλό είναι να δημιουργούμε πλεονάσματα. Και αυτή η δεκαετία του 1990 που ήταν καλή για την Ευρώπη θα μπορούσε να ε, είχε δημιουργήσει πλεονάσματα στο δημοσίο και στον ιδιωτικό τομέα και τώρα θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη θέση. αυτά και σας ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Ε, βεβαίως όσο ο Υπουργός Οικονομίας μπορεί να έχουμε κάποια προκατάληψη γιατί ξέρετε πριν από 10 χρόνια στην Ουγγαρία είχαμε εφαρμόσει ένα σχέδιο εθνικής ανάπτυξης και η ουσία της επιτυχίας του σχεδίου ήταν πως δώσαμε οξυγόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιδοτήσεις και τους επιτρέψαμε να κάνουν κεφαλαιακές επενδύσεις και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Γιατί όπως ξέρετε 70% των θέσεων εργασίας του ιδιωτικού τομέα στην Ουγγαρία είναι σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οπότε νομίζω πως η στρατηγική του 2020 έχει τους σωστούς στόχους, την αύξηση δηλαδή της απασχόλησης, ε, εκπαίδευση, πρέπει να ενισχυθεί και αυτό βεβαίω εξυπηρετείται και εξυπηρετήθηκε και από το σχέδιο τότε Ευχαριστώ. Καταφέραμε να βολέψουμε 14 ερωτήσεις. Ελπίζουμε και προσβλέπουμε στο να συναντηθούμε και πάλι προς το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Εγώ δεν μπορώ να ψέξω την Ουγγρική Προεδρία για το γεγονός ότι προσπαθεί να κάνει συναντήσεις σε ψηλό επίπεδο και νομίζω ότι με τον ενθουσιασμό αυτό μπορούμε να συνεργαστούμε και οι δύο πλευρές με πολύ καλό τρόπο και προσβλέπω λοιπόν στο να πραγματοποιηθούν οι στόχοι σας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, λέει ο υπουργό. If you just, uh, just have a couple of minutes break. Δύο λεφτά διακοπή για να αποχαιρετήσω τον κύριο Υπουργό γιατί θα έρθουν και άλλοι εισηγητές. Λοιπόν, επανερχόμαστε. Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο από την επόμενη συζήτηση που επίκειται. Έξι εκθέσεις πρέπει να συζητήσουμε για τα θέματα οικονομικής διακυβέρνησης που εμπλέκονται στη δέσμη αυτή. Καθίστε λοιπόν παρακαλώ. Θα κάνουμε μια κοινή συζήτηση στα σημεία 4, 5, 6, 7, και 8. Και θα ακολουθήσουν οι συγητές με αυτή τη σειρά. Με τη σειρά που αναφέρονται, κυρία Βόρτμαν Κόλ, Φέο, Φερέιρα, Γκουλάρ, Χάγκλαντ και τέλος και η κυρία Φόρτ. Αν θέλετε λοιπόν να καθίσετε και να ηρεμήσετε, δίνω το λόγο καταρχήν στην κυρία Βόρτμαν Κόλ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος όλων των εισηγητών λέγοντας ότι προφανώς με μεγάλη προσδοκία πλησιάζουμε αυτή τη στιγμή της πρώτης συζήτησης στην Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή για τα σχέδια εκθέσεων που εμπλέκονται στο πακέτο αυτό για την οικονομική διακυβέρνηση. Οι εκθέσει αυτέ έχουν συνταχθεί εν συνεργασία. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια να συναντηθούμε μεταξύ μας, να συζητήσουμε μεταξύ μα τι ακριβώς θα έπρεπε να είναι η θέση η οποία θα παρουσιαστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ποια θα ήταν η καλύτερη θέση για το Κοινοβούλιο. <clears throat> και όπως σας είπα προσβλέπω στη συνέχιση του έργου μας με έναν τρόπο ανοιχτό και επικοδομητικό, όχι μόνο με τους συζητητές αλλά και με όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Είναι απαραίτητο να συνεργαστούμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια στεναρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εναντίον του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Σα υπενθυμίζω ότι αυτό δεν είναι μονάχα ένα από τα πιο σημαντικά νομοθετικά πακέτα σε αυτήν την ε, θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συγχρόνως είναι και η πρώτη φορά που εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δρούμε ως συν για τέσσερις από τις έξι εκθέσεις του πακέτου. Προσπαθήσαμε λοιπόν να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, ώστε οι έξι αυτές προτάσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ως δέσμοι, ως σύνολο. Και το Κοινοβούλιο δεν πρέπει απλώς να είναι παρόν στις εκθέσεις που είναι <clears throat> με ίσα δικαιώματα συνομοθέτης, αλλά και στις έξι εκθέσεις. Και μπορούμε να διαγράψουμε <clears throat> μια εντολή διαπραγμάτευση ούτω ή από την πλευρά του Κοινοβουλίου, μόνο όταν έχουμε περάσει μια πρώτη εξέταση των εκθέσεων αυτών και έχουμε καθορίσει την πορεία πλευσεώς μας. Όπως φάνηκε και από τη συζήτηση με τον Ούγγρο Υπουργό, ο στόχο είναι να περατωθεί η εξέταση του πακέτου τον Ιούνιο. Αυτό όμω εξαρτάται και από τη στάση που θα κρατήσει το Συμβούλιο, το κατά πόσο το Συμβούλιο θα δείξει ανοιχτό πνεύμα για να λάβει υπόψη τι θέσει τι οποίε θα προτάξει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό είναι το μόνο έδαφο στο οποίο μπορούμε να επιτύχουμε μια κοινή λύση τον Ιούνιο. Ω εισηγητέ, εμεί προσπαθήσαμε να βρούμε σύμπτωση απόψεων για κέρια θέματα. Συγχρόνως όμως θα πρέπει να επεξεργαστούμε περισσότερο το πώς αυτή η προσέγγιση θα μεταφραστεί συγκεκριμένα σε κάθε ένα από τα νομοθετικά ε, νομοθετήματα που έχουμε ενώπιόν μας. Τέσσερα στοιχεία αυτής της κοινή προσέγγισης θέλω να αναφέρω και τον τρόπο με τον οποίο τη συμπεριέλαβα στη δική μου έκθεση για το προληπτικό σκέλος της, ε, και την εποπτεία των οικονομικών πολιτικών. Καταρχήν θέλουμε ένα ισχυρό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να αποφύγουμε να υπόκεινται όλες οι κρίσεις και οι αποφάσεις σε πολιτικό παζάρι μεταξύ των κρατών μελών στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλοι ξέρουμε τι προέκυψε από αυτά τα αλογοπάζαρα τα προηγούμενα χρόνια. Γι' αυτό θέλουμε να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να ακολουθηθεί η κοινοτική μέθοδος. Στην έκθεσή μου εγώ επίσης ζητώ να υπάρξει ταχαίως η χρήση της ε, ψηφοφορίας με ειδική πλειοψηφία στη σχέση, σε σχέση με την εφαρμογή του προληπτικού σχέλους εποπτείας. Και δεύτερον, σε όλες τις εκθέσεις θα βρείτε τα στοιχεία μιας εργαλειοθήκης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία αυτά ήδη σε ένα πρώιμο επίπεδο. Εγώ στη δική μου έκθεση τονίζω την ανάγκη να υπάρχουν αυξημένες απαιτήσει αναφορών και εκθέσεων όταν υπάρχει μια απόκληση των κρατών μελών από τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί σε μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό επίπεδο. Επίσης αύξηση της εντολής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ενδεχομένως Καλύτερη ποιότητα και μεγαλύτερη χρήση στατιστικών στοιχείων και με όλο αυτόν τον τρόπο προσπαθώ πράγματι να ενισχύσω το προληπτικό σκέλο τη εποπτεία, γιατί ο καλύτερο τρόπο να αποφύγουμε τι κυρώσει είναι να είναι ισχυρή και στεναρή η προληπτική διαδικασία εποπτείας σε ένα πρώιμο επίπεδο και επομένω έτσι μπορεί να αποφύγει κανεί προσαρμογέ, οι οποίε μπορούν να είναι οδυνηρές όταν έχει ήδη δημιουργηθεί υπερβολικό χρέο ή δημοσιονομικό έλλειμμα. Το τρίτο στοιχείο που θέλω να τονίσω είναι ότι με το πακέτο αυτό ο στόχος μας να επιτύχουμε ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες μας. Γι' αυτό πρέπει να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών και την κοινωνική σταθερότητά τους. Για να γίνει κάτι τέτοιο, η βάση, το θεμέλιο μας <clears throat> θα πρέπει να είναι υγιείς δημοσιονομικές πολιτικές σε σχέση και με το χρέος και με το δημοσιονομικό έλλειμμα, όπως λέει η εκθεσή μου. Αλλά και αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ισχυρή μακροοικονομική εποπτεία και θετική οικονομική διακυβέρνηση της στρατηγικής Ευρώπη 2020. Ξέρουμε πως το παρόν αυτό είναι σχετικά ισχνό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτή την πτυχή, γιατί και αυτή όπως είπα είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προλάβουμε σημαντικά προβλήματα στο μέλλον, εγώ συμπεριέλαβα στην εκθεσή μου και τα ευρωπαϊκά εξάμεινα στο νομοθετικό κείμενο, όχι μονάχα για να εξασφαλίσει ότι υπάρχει δέσμευση από τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν την επίτευξη των στόχων για υγεία δημόσια οικονομικά και οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης και για να τονίσω περισσότερο το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων στη σύνολη αυτή διαδικασία. <clears throat> Μια στεναρή διαδικασία λοιπόν εποπτείας, όχι μόνο στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά στην γενικότερη ε, στρατηγική μακροοικονομικής εποπτείας και τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Όχι μόνο το Εθνικό, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα πρέπει να συμμετέχουν και φυσικά και οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει να διαδραματίσουν ένα ρόλο και αυτό να εξασφαλιστεί. Και αυτό βρίσκεται μέσα στην έκθεσή μου. Τέταρτο στοιχείο είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε τη λεγόμενη οικειοποίηση, ownership σε εθνικό επίπεδο. Είναι απαραίτητο από την άποψη η οικονομική διακυβέρνηση να είναι κάτι το οποίο θα αφορά όλους και θα είναι ζήτημα κοινή ευθύνη των κρατών μελών και των εθνικών κοινοβουλίων. Προς το παρόν βλέπουμε πάρα πολλά που έχουν να κάνουν με διοικητικέ διαδικασίες, προετοιμασία προγραμμάτων σταθερότητας, σύγκληση, εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεως κτλ. τα οποία αποστέλλονται στις Βρυξέλλες αλλά <clears throat> από την άλλη πλευρά οι εθνικές κυβερνήσεις λειτουργούν αυτόνομα σε ό,τι αφορά την εκπόνηση προϋπολογισμών στα εθνικά κοινοβούλια και δεν υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των δύο διαδικασιών. Γι' αυτό εγώ συμπεριέλαβα στην εκθεσή μου την ανάγκη να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και των κοινοβουλίων <clears throat> για την εκπόνηση και την έγκριση των προγραμμάτων στα, σταθερότητας και ανεξάρτητες στατιστικές προβλέψεις, ώστε να γίνεται καλύτερη συζήτηση στα κράτη-μέλη και στα κοινοβούλια. Η έκθεσή μου προτείνει επίσης να ενσωματώσουμε στην εθνική νομοθεσία τους στόχους του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη. Ξέρω ότι αυτό μπορεί να είναι αμφιλεγόμενο, να οδηγήσει σε συζητήσεις, αλλά προσβλέπω σε τέτοιου είδου συζητήσει γιατί νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη δέσμευση από την πλευρά των κρατών μελών για την επίτευξη των στόχων του Συμφώνου. Είναι σαφέ και αυτό φαίνεται και από τον τρόπο που όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να περάσουν σε συγκεκριμένε νομοθετικέ ρυθμίσει, ότι εμεί ω Κοινοβούλιο χρειάζεται να επεξεργαστούμε περισσότερο αυτά τα νομοθετήματα. Ένα από τα κέρια επίση θέματα σε ό,τι αφορά την προληπτική εποπτεία είναι η επίτευξη μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων. Συζητήσαμε αυτό το ζήτημα διαμακρών στο παρελθόν και επίσης το θέμα της σόφρονος λήψης αποφάσεων σε σχέση με τη χάραξη πολιτικής το σημείο αυτό εγώ δεν το έχω τροποποιήσει, αλλά εγώ είμαι έτοιμη να συζητήσουμε περισσότερο για περαιτέρω διευκρίνηση στο σημείο αυτό. Είναι απαραίτητο τα κράτη-μέλη να <clears throat> ακολουθήσουν συγκεκριμένες πορείες και μονοπάτια προσαρμογής προς την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων, που δεν είναι ευρωπαϊκού τύπου ρετσέτες ή ηλιοτυπίες, αλλά πρέπει να είναι τα δικά τους σχέδια και οι του τους στόχοι σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο των κρατών μελών δηλαδή. Τονίζω περισσότερο στο κείμενο ότι δεν πρέπει να υπάρξει η αξιολόγηση μονάχα του προφίλ του χρέους και του επίπεδου του χρέους, αλλά επίσης και του προβλήματος της βιωσιμότητας των δημοσίων οικονομικών. Και αυτή η πτυχή πρέπει να ληφθεί υπόψη. Είχαμε επίσης συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κατά την άποψη της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας υπάρχει ιδιαίτερα μεγάλο περιθώριο ελιγμών για τα κράτη-μέλη μέσα σε αυτή την οδηγία, ώστε να μην είναι υποχρεωμένα να συμμορφώνονται απόλυτα με τα κριτήρια για το χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα. Εγώ δεν πείραξα όμω αυτή τη διατύπωση τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το περιθώριο ελιγμών, γιατί πιστεύω ότι σε ορισμένε περιπτώσει πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι κρίσει των κρατών μελών σε σχέση με το γενικό στόχο. Παραδείγματο χάρη σε εποχέ σοβαρή οικονομική κάμψη, τότε η δυνατότητα να ακολουθήσουν τους δικούς τους δρόμους στα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να γίνει αποδεκτή. Ένα άλλο θέμα το οποίο αξίζει να συζητηθεί είναι το πώς θα μπορέσουμε να συνεκτιμήσουμε επενδύσεις, τις επενδύσεις των κρατών μελών. Και εδώ πάλι άφησα άθικτο το κείμενο της Κομισιόν, γιατί το κείμενο της Κομισιόν λέει ήδη ότι όταν καθορίσουμε την πορεία προσαρμογής, την τροχιά προσαρμογής, η εφαρμογή μιζώνων μεταρρυθμιστικών μεταρρυθμίσεων που μπορούν να αυξήσουν το δυναμικό για ανάπτυξη και μπορούν να έχουν επαληθεύσιμο αντίκτυπο στην μακροχρόνια ε, βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών πρέπει να ληφθούν υπόψη. Και εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη. Επομένω, άφησα αναλύωτο το κείμενο τη Κομισιόν για το θέμα αυτό. Εγώ προσλέπω σε μια περαιτέρω συζήτηση για τα θέματα αυτά πιστεύω προς το παρόν ότι δεν έχω να πω τίποτα περαιτέρω και θέλω επίσης να υπογραμμίσω, τελευταίο αλλά όχι ότι εγώ <clears throat> έχω εστιάσει την προσοχή μου σε αυτό το νομοθετικό πακέτο. Συγχρόνως έχω απόλυτη επίγνωση ότι αυτό είναι μονάχα ένα πετραδάκι, μία ψηφίδα μονάχα στο σύνολο του πακέτου προτάσεων που πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως εργαλείο αντιμετώπισης της κρίσης. Επίση ο μηχανισμό αντιμετώπισης των κρίσεων. Οι αλλαγές της συνθήκης και ίσως άλλες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και να συνεξεταστούν. Αλλά είναι μια σημαντική ψηφίδα στο μοσαϊκό η πρόταση αυτή που ανέφερα το να αυξήσουμε την προληπτική εποπτεία και επομένως βλέπω και στα σχόλιά σας και την περαιτέρω συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ λέει και η πρόεδρος, ο κύριος Φέιου. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το να ευχαριστήσω όλους για τη βοήθεια που μου έχουν δώσει, τη γραμματεία συγκεκριμένα της Επιτροπής μας, η οποία έκανε δυνατό να παρουσιαστεί σε αυτή τη χρονική στιγμή η έκθεσή μου. Η έκθεση, η οποία είναι μία από τις έξι εκθέσεις που ανέφερε η κυρία Βόρτμαν Κόλ, έχει μεγάλη σημασία αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί βρισκόμαστε σε μια συγκυρία που μας υποχρεώνει να εξεύρουμε θεσμικού χαρακτήρα μηχανισμούς για να υπερβούμε την κρίση, αλλά όχι μόνο, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και να εμποδίσουμε μελλοντικέ κρίσεις. Η έκθεσή μου έχει ως ειδικό αντικείμενο την διορθωτική πτυχή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω εδώ είναι ότι η έκθεση αυτή περιορίζει τον εαυτό της σε μία σειρά θέματα λόγω και των διατάξεων της ε, συνθήκης Λισαβόνας που δεν αφήνουν πολύ περιθώριο στο παράγωγο δίκαιο. Καταρχήν, αυτό το οποίο επιζητεί είναι να υπάρχει μία καλύτερη μορφή λειτουργικού καθορισμού του τι είναι το υπερβολικό έλλειμμα μέσα στη διαδικασία υπερβολικού έλλειμματος. Δηλαδή, για την χρηματοοικονομική σταθερότητα της ζώνης του ευρώ και των άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μονάχα το δημοσιονομικό έλλειμμα αλλά και το συνολικό χρέος. Η τροποποίηση εδώ που έχω κάνει σε σχέση με το κείμενο της Κομισιόν είναι η εξή. Σε σχέση με τον κανόνα για τη μείωση του χρέους κατά ένα εικοστό το χρόνο. Η Κομισιόν είχε προτείνει αρχικά ότι μέχρι να φτάσουμε το 60% του δημοσίου χρέους θα έπρεπε να ήταν το 10, το 1 δέκατο το χρόνο. Η ίδια αρχή εφαρμόζεται τώρα και από την Κομισιόν και από εμάς. Εμείς μιλάμε για ένα 20 μέσα στα πλαίσια τριετούς χρονικής περίοδου. Ξέρω ότι αυτό είναι τώρα μια πρόταση η οποία είναι αμφιλεγόμενη ενδεχομένως, μπορεί να δημιουργήσει ε, διαφωνίες γιατί έχουμε να κάνουμε με διαφορετικούς κανόνες και ενδεχομένως υπάρχει το θέμα του της αυστηρότητα του κριτηρίου αυτού σε σχέση με αυτό που έλεγε η Κομισιόν. Ε, επίσης, θα πρέπει κατά την άποψή μου να μειωθούν οι προθεσμίες σε σχέση με την παράδοση των ε, στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη συνεκτίμηση της κατάστασης, ώστε όταν περάσουμε στη φάση η οποία είναι η διορθωτική φάση βάσει του Συμφώνου Σταθερότητας, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να μειωθεί και να συμπιεστεί στο ελάχιστο ο χρόνος για τον οποίο βρίσκεται ένα κράτο σε κατάσταση δυσκολία. Τρίτο σημείο το οποίο θέλω να υπογραμμίσω, η έκθεση αυτή, όπως και σε άλλες εκθέσεις, προτείνει οι κυρώσει να πληρώνονται όχι μόνο για τα κράτη-μέλη τα οποία προς τα κράτη που έχουν ε, καλή χρηματοοικονομική κατάσταση, αλλά προς τα ταμεία τα οποία έχουν σαν στόχο να ενισχύσουν τη σταθερότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέταρτον. Ένα από τα αμφιλεγόμενα στοιχεία αυτού του νομοθετήματος και της εκθεσής μου είναι το να αντιμετωπιστεί το κόστος των συνταξιοδοτικών ταμείων μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας για το υπερβολικό χρέος ή έλλειμμα στις συζητήσεις που γίνονται τώρα στην ομάδα των 14, ο στόχος είναι να υπάρχουν ορισμένες άλλες μορφές ε, δαπανών οι οποίες δεν θα εμπίπτουν στη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. Αλλά εγώ εδώ έχω παραμείνει πιστός στην αρχική πρόταση της Κομισιόν. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία μια μεγαλύτερη συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία αυτή όπω και στι άλλε εκθέσει. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αυτή θα πρέπει να υπάρξει δυνατότητα δημόσιου διαλόγου και η δυνατότητα να κληθούν οι αρμόδιες επιτροπές για την εφαρμογή του Συμφώνου σταθερότητα στα κράτη-μέλη για να εξηγήσουν καλύτερα, μάλλον να προσκληθούν τα κράτη-μέλη σε αυτές τις επιτροπές για να εξηγήσουν καλύτερα την θέση τους σε σχέση με τα ζητήματα προπολογισμού. Όπως έλεγα προηγουμένως στους συναδέλφους, τα σημεία τα οποία είναι τα πιο ε, επίμαχα είναι ακριβώς ο ρυθμός της μείωσης του χρέους κατά 0,5% ένα διακοσιωστό μάλλον και όχι το 20 που έλεγχε προηγουμένως λαθασμένα αντί για ένα εκατοστό. Κάτι ακόμα το οποίο θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι αυτό είναι μονάχα ένα κομμάτι μιας συνολικής διαδικασίας που έχει να κάνει με την οικονομική διακυβέρνηση. Συζητούμε εδώ το Σύμφωνο Σταθερότητος και Ανάπτυξης. Έχουμε να συμπεριλάβουμε και το θέμα της αντιμετώπισης των, δημοσιο... μακροοικονομικών ε, ανισοτήτων, αλλά είναι απαραίτητο σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση να μπορούμε να έχουμε μια κοινή αντιμετώπιση. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην τωρινή συζήτηση, αλλά είναι σημαντικά, όπως είναι τα λεγόμενα ομόλογα project, ομόλογα σχεδίων που παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Κομισιόν ή ακόμα και υπενθυμίζω τη συζήτηση που έγινε μεταξύ των έξι εισηγητών και εδώ στην Επιτροπή μας μετά από μία σειρά ακροάσεων <clears throat> και που συνάπτεται με τα ευρωομόλογα και όπου είναι φανερό ότι δεν υπάρχει ενιαία θέση μεταξύ των κοινοβουλευτικών πολιτικών ομάδων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να κινηθούμε προ μια κατεύθυνση η οποία θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη θεσμικοποίηση των θεμάτων αυτών. Είναι απαραίτητο να δώσουμε πολιτικέ απαντήσει σε προβλήματα τα οποία είναι οικονομικού χαρακτήρα αν θέλετε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ στο οικονομικό επίπεδο, αλλά δεν έχει ακολουθήσει η πολιτική Είναι, ένωση. είναι μια στιγμή να τροποποιήσουμε αυτή την ισορροπία. Είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρέμβαση. Είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου και λειτουργία, ώστε να αντιμετωπιστούν και όλες αυτές οι απαραίτητες διαφορετικές αλλαγές που γίνονται στα κράτη-μέλη και οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε το σύμφωνο σταθερότητος να είναι σύγχρονο στην πραγματικότητα και στην πράξη και σύμφωνο ανάπτυξης. Συμφων... Συζητούμε λοιπόν σήμερα τα θέματα αυτά της οικονομικής διακυβέρνησης <clears throat> και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά κράτη τα οποία δεν έχουν προβεί στις απαραίτητες διαφορετικές αλλαγές που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη των οικονομιών τους. Κλείνω με δύο ακόμα παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αυτό με ικανοποιεί ιδιαίτερα, έχει δείξει μεγάλη ενεργητικότητα και ενδιαφέρον για το θέμα αυτό. Έχει ήδη ως θεσμικός φορέας δώσει την άποψή του με μια προηγούμενη έκθεση. Συζητά τώρα τις έξι εκθέσεις που αναφέραμε και γι' αυτό εγώ βρίσκω ακατανόητο που Πολλέ φορέ το Συμβούλιο δεν αναφέρεται καθόλου στη θέση του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι κατά τη διάρκεια τη διαδικασία αυτή το Συμβούλιο θα αράξει πορεία πλεύση και ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατό να μπορέσουμε να συζητήσουμε από κοινού τι έξι αυτέ εκθέσεις, παρά το γεγονός ότι τέσσερι είναι σε διαδικασία συναπόφαση και δύο όχι, είναι απαραίτητο όμω να συνεχίσουμε την παραλληλία τη συζήτηση αυτών των εκθέσεων, ώστε μέχρι το τέλο τη διαδικασία που ελπίζω να είναι το καλοκαίρι, να υπάρξει μια συνολική συζήτηση και των έξι εκθέσεων όμου. Ευχαριστώ πολύ και προσδοκώ να ακούσω και τις συμβολές των συναδέλφων για το θέμα αυτό. Thank you very much. Um, Elisa. Η κυρία Φερέιρα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ είμαι η συγγήτρια για την έκθεση που αφορά τις μακροοικονομικές ανισορροπίες και όπως και οι προλαλήσαντες συνάδελφοι, εγώ θα ήθελα να σας αναφέρω ότι το νομοθετικό αυτό πακέτο, το οποίο έχει παρουσιαστεί από την Κομισιόν στις 29 Σεπτεμβρίου του 2010, είναι ένα πολύ σημαντικό πακέτο, χωρίς καμία αμφιβολία, για να μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της Ευρώπης και του, του ίδιου του ευρώ. Για μας η μεγάλη πρόκληση ενώπιόν μας είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ μιας δημοσιονομικής πειθαρχίας συγγνώμη, που να είναι βιώσιμη και αηφόρα και πολιτικές δημοσιονομικές αυτού του χαρακτήρα αφενός, αλλά από την άλλη πλευρά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και μια συνεκτικότητα μεταξύ αυτής της αντιμετώπισης και της ανάγκης να δημιουργήσουμε απασχόληση, ανάπτυξη και σύγκληση στα οικονομικά μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο κατευθύνσεις οι οποίες θα πρέπει να συνδυαστούν με σωστό τρόπο μέσα στη στρατηγική που θα ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δική μου πολιτική ομάδα, και που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συγκλίνει στην θέληση και την αναγκαιότητα να συνεργαστεί με τις άλλες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για μια κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αλλά το πακέτο που έχουμε στα χέρια μας θα έχει μονάχα νόημα αν εφαρμοστούν με σωστό τρόπο όλες οι διατάξεις του και επίσης αν εξασφαλιστεί η συμπερίληψη δύο ακόμα πτυχών. Από τη μία πλευρά είναι απαραίτητο το πακέτο της μακροοικονομικής διακυβέρνησης να μην περιοριστεί στο να εφαρμόζει κυρώσεις στους παραβάτες. Θα πρέπει να δημιουργήσει ισχυρούς μηχανισμούς αλληλεγγύης, ώστε να επιτρέψει τη σωστή λειτουργία της ζώνης του ευρώ. Γι' αυτό η καλύτερη εξέταση των θεμάτων των ευρωομολόγων και ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου που δεν θα είναι μόνο διακυβερνητικό αλλά ενωσιακό, κοινοτικό, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Επομένως, η διάσταση της ανάπτυξης και της δημιουργίας απασχόλησης και η εξασφάλιση της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής δεν μπορούν να παραμείνουν σε επίπεδο μονάχα ασαφών δηλώσεων. Η λειτουργία του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα πρέπει να επιτρέψει με τρόπο βιώσιμο να υπάρχει ανάπτυξη σύγκληση, ενώ συγχρόνως επιτυγχάνονται οι στόχοι της εξυγίανσης των δημοσίων οικονομικών. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο, αυτή η ισορροπία δεν θα μπορέσει να είναι βιώσιμη και να έχει αηφόρο χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε και προς μια άλλη διάσταση που είναι η συνολική χρέωση ενός κράτους μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020 για να προχωρήσουμε στις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα και έχουμε ήδη εργαστεί προς την αυτή την κατεύθυνση να εξασφαλίσουμε ότι το έργο των εισηγητών και το έργο των πολιτικών ομάδων θα οδηγήσει σε μια στεναρή κοινή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. <clears throat> Γιατί έχουμε απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι οι πολίτες προσδοκούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να τους δώσει μια απάντηση που να έχει αυτά τα οδηγά στοιχεία ενώπιον της μεγαλύτερης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που έχει γνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από την δημιουργία της και ιδίως από τη στιγμή που υιοθέτησε το ενιαίο νόμισμα. Γι' αυτό πρέπει να δείξουμε απόλυτη δέσμευση για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα επιτύχει του στόχου τη και επίση για να εξασφαλίσουμε ότι τα έξι αυτά νομοθετικά κείμενα τα οποία ε, εξετάσουμε θα έχουν απόλυτη εσωτερική συνοχή. Όπω είπαν και οι συνάδελφοι, νομίζω ότι έχουμε πετύχει ένα λογικό βαθμό σύγκληση μεταξύ των εξή ηγητών και ελπίζουμε θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε προ την κατεύθυνση αυτή για να επιτύχουμε βελτιώσει σε μια σειρά θεμάτων στα οποία έχουμε ήδη μια καταρχήν σύγκληση απόψε. Ιδίω έχουμε επιτύχει σύγκληση για τα θέματα της βελτίωσης της δημοκρατικής νομιμοποίησης με την ε, συμμετοχή και άλλων εμπλεκομένων και φορέων, stakeholders, με την συμμετοχή των Εθνικών Κοινοβουλίων επίσης και όχι μόνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επίσης κάτι σημαντικό να μπορέσουμε να δώσουμε πραγματικό περιεχόμενο στη στρατηγική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης και να χρησιμοποιήσουμε με έναν τρόπο ευφυή και σοβαρό και φυσικά και σωστό τον χώρο ο οποίος δημιουργείται, το χώρο παρέμβασης που δημιουργείται από το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Εγώ είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη ε, από αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες, οι οποίοι τόνισαν και πάλι ότι υπάρχει απόλυτα ανοιχτό πνεύμα για θέματα που για μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Παραδείγματο χάρη, ο συνδυασμό των στόχων σε σχέση με το χρέο και με το δημοσιονομικό έλλειμμα που κατά την άποψή μας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με τρόπο ο οποίος είναι αυτόματος, αλλά θα πρέπει να είναι αντικείμενο μιας διαδικασίας διαπραγματεύσεων με το εμπλεκόμενο κράτος μέλος, μιας διαπραγμάτευσης η οποία να είναι συνεκτική με την επίτευξη των μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων αυτού του κράτους μέλους και μόνο έτσι μπορεί να καθοριστούν οι στόχοι για το χρέος και για το έλλειμμα, όχι με μηχανιστικέ και απόλυτε αριθμητικές τιμέ που δεν έχουν κανένα νόημα. Επίση, χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε ότι υπάρχει ανοιχτό πνεύμα για να συζητηθεί και η έννοια τη φρόνιμη, ισόφρονο δημοσιονομική πολιτική, η οποία επιτυγχάνει την βιωσιμότητα σε οικονομικό και δημοσιονομικό επίπεδο. Ένα τρίτο σημείο είναι το να αντιμετωπιστούν οι επενδύσεις που έχουν να κάνουν με την μεταρρύθμιση των, δημοσι... των ε, συστημάτων μαζί με άλλες ε, επενδύσεις οι οποίες είναι σημαντικές για την προώθηση της ε, ανάπτυξης όπως είναι οι επενδύσεις στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση κτλ. Πρέπει να είναι από κοινού λοιπόν η αντιμετώπιση αυτών των ε, επενδύσεων και με τον τρόπο αυτό ελπίζουμε θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε περισσότερη σύγκληση απόψεων. Τέλος, το κείμενο για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες τονίζει ότι αυτό είναι το μόνο εργαλείο μέσα στο πακέτο όπου είναι δυνατόν να υλοποιήσουμε τον προληπτικό χαρακτήρα της παρέμβασης του Συμφώνου Σταθερότητας. Το οποίο σημαίνει ότι όχι μόνο βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες να μπορούμε να διακρίνουμε, αλλά και αυτές οι οποίες μπορούν να είναι οι εύθραστες πηγές μιας πορείας σύγκλησης, οι οποίες όταν επαναλαμβάνονται επί σειρά ετών αντανακλούν πραγματικά διαφορετικά προβλήματα, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε αυξανόμενες ε, αποκλίσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως μέσα στο, στη ζώνη του ευρώ, όπως φάνηκε στην τελευταία δεκαετία. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, εμείς Θέλουμε και πρέπει να βρούμε ένα τρόπο με τον οποίο θα υπάρχει και κάποια συμφωνία για τις δράσεις οι οποίες γίνονται από ένα κράτος αλλά έχουν αποτελέσματα και σε άλλες χώρες. Το λεγόμενο spillover effect στα αγγλικά. Δηλαδή το γεγονός ότι ξεπερνούν τα εθνικά όρια πολλές φορές οι αντίκτυποι αυτών των δράσεων. Το λεγόμενο βαθμολόγιο, το scoreboard, το οποίο είναι σε κατασκευή αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει χωρίς την ενεργή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πρέπει μέσα από μια συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και της Κομισιόν, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να σταθμίσουμε μια σειρά από που καταδεικνύουν όχι μονάχα τις εσωτερικές ανισορροπίες αλλά και τις εξωτερικές ανισορροπίες αλλά και την χρονική διάσταση, ιδίως τη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, που ξεπερνάει μια απλώς συγκυριακή και ονομαστική αξιολόγηση. Πρέπει να έχουμε μέγιστους και ελάχιστους δείκτες, να καθορίσουμε τέτοιου είδου δείκτες, αλλά πιστεύω ως εισηγήτρια ότι το βαθμολόγιο δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται με αυτόματο και μηχανιστικό τρόπο. Θα πρέπει να είναι ένας τρόπος να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνοδεύεται το βαθμολόγιο με επιτόπιες ε, αποστολές οι οποίες θα πληροφορούν τα αρμόδια κράτη-μέλη και την Κομισιόν για, το, για τη φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζονται και για την καλύτερη τροχιά βελτίωσης και διόρθωσης αυτών των προβλημάτων. Αυτό θα πρέπει να είναι μια φυσιολογική διαδικασία και όχι μια διαδικασία η οποία θα λαμβάνει χώρα μονάχα σε καταστάσεις κρίσης. Και υπάρχει και απόλυτη συμφωνία μεταξύ εμού της Ιδίας και του εισηγητή που έχει να κάνει με τις κυρώσεις για το νόημα των κυρώσεων και θα τα παρουσιάσει καλύτερα φυσικά συναδελφός μου γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ιδίως σε αυτό το τομέα οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται να χειρώνουν την έλλειψη θέλησης δράσης και όχι την αδυναμία δράσης όταν οι μακροοικονομικές ανισορροπίες είναι τόσο πολύπλοκες και ιδίως είναι τόσο, τόσο δύσκολο να μπορέσει να καταλογίσει κανείς τις αιτίε αυτών των ανισορροπιών σε συγκεκριμένες δράσεις μιας και μόνο χώρας. Επομένως πρέπει να ληφθεί υπόψη το σύνολο αυτών των πτυχών. Τέλος είναι απαραίτητο αυτή η εργασία. Και η λειτουργία σε όλο αυτό το πλαίσιο αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών να συνδέεται και να συσχετίζεται πάρα πολύ στενά με το έργο το οποίο γίνεται σε σχέση με τη ρύθμιση των αγορών και την εποπτεία των αγορών και όλος ιδιαίτερος σε σχέση με το Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε πραγματικά να υπάρχει ε, ουσιαστικά και αμοιβαία εκμετάλλευση από τις δύο πτυχές και από τις φορείς αυτούς, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα και της, του προβλήματος και τις ενδεχόμενες ανισορροπίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν, εάν δεν υπάρχει συντονισμός. Όλα αυτά λοιπόν έχουν νόημα όταν υπάρχει μια σωστή άρθρωση με μια επαναθέρμανση της πορείας προς την σύγκληση των κρατών μελών και εκεί περιμένουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Σίλβη. Ευχαριστώ πολύ Σάρων. Σας ευχαριστώ όλους σας. Πολλά είπαν οι συνάδελφοι και συμφωνώ με το γενικό αυτό αίσθημα ότι δηλαδή ε, προσπαθήσαμε όλοι να συνεργαστούμε όσο πιο καλά γίνεται και όλοι μας θέλουμε να κάνουμε έκκληση αυτή, αυτές η εργασία να πάει πέραν των εισηγητών μια, να είναι μια εργασία της Επιτροπής μας, γιατί έχουμε σημαντική ευθύνη. Σας θυμίζω ότι για πρώτη φορά το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει τη δυνατότητα να είναι συνομοθέτης για το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης που την πρώτη φορά το διαπραγματεύτηκαν χωρίς το Κοινοβούλιο. Το μεταρρύθμισαν μετά χωρίς το Κοινοβούλιο. Πολιτικό μήνυμα λοιπόν. Όλοι μαζί θα πετύχουμε να επιβάλλουμε ορισμένες απόψει στο Συμβούλιο. Διαφορετικά ο κίνδυνο είναι να χάσουμε όλοι μα. Δεν μπορεί μία ομάδα να ωφεληθεί μόνη της από το εγχείρημα αυτό. Θα ήταν κάτι πολύ βραχυπρόθεσμο αυτό. Έπειτα το μήνυμα προς τον πολίτη θέλουμε να είναι θετικό. Ίσως να είμαι υπερβολικά αφελής και αισιόδοξη. Ένα θετικό της κρίσης είναι ότι μας δείχνει τι δεν πήγαινε καλά στην Ευρωζώνη και πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να διορθωθεί. το θέμα σύγκλησης που αναφέρθηκε και επαναλαμβάνω ότι συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν, είναι αυτό που είπε η Κορίν. Καλύτερη πρόληψη. Εγώ ασχολούμαι με τι κυρώσει. Μακάρι να μην χρειαστεί να εφαρμοστεί το κείμενό μου. Μακάρι να χρειάζεται, μακάρι να πετυχαίνουμε πρόληψη και χωρί κυρώσει. Δεύτερον, να συμπεριληφθεί το χρέο παράλληλα με το έλλειμμα. Αυτό υπήρχε στο κείμενο. Δυστυχώ, όπω είπε ο Ιούγκο, κάπω υποτιμήσαμε το σημείο αυτό όχι να βγούμε από την κατάσταση της υπερχρέωσης στην οποία βρισκόμασταν. Αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε και άλλο θέμα, δεν έχω αντίρρηση, δεδομένου ότι για όλα τα θέματα πρέπει να κάνουμε την προσπάθεια να πετύχουμε ισορροπία μεταξύ του είμαστε από τη μια μεριά έξυπνοι και ελαφροί, ευκίνητοι, από την άλλη μεριά η πειθαρχία να παραμείνει. Το κείμενο της Λίζα για τις μακροοικονομικές ε, ανισομέρειες και αυτό είναι σημαντικό, γιατί για πρώτη φορά προσπαθούμε να έχουμε εργαλεία που να, είναι, να μην είναι πολύ χοντροκομμένα. Το δημόσιο χρέος, το δημόσιο έλλειμμα, αλλά βλέπουμε ότι η κρίση μας έδειξε ότι σε ορισμένε χώρες υπάρχουν προβλήματα και όσον αφορά την ιδιωτική δαπάνη και κατανάλωση. Και υπάρχει μια απόκληση, αποκλήσεις μάλλον μέσα στη νευροζώνη. πολύ οικονομολόγοι το επεσήμεναν αυτό, έχουμε ένα σύστημα που αντί να οδηγήσει σύγκληση μπορεί να οδηγήσει απόκληση. Πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη της οικονομίας και να βάλουμε μέσα και τα λεγόμενα spillover στα αγγλικά. Να πάψει να υπάρχει αυτή η συνολική δυσπιστία ή αδιαφορία μάλλον. Δηλαδή ο καθένα έλεγε Α, έχουμε ένα νόμισμα, ο καθένα κοιτάει τα δικά του, αδιαφορούμε τι γίνεται στην αυλή του γείτονα. Δεν γίνεται αυτό πια. Στο Κοινοβούλιο λοιπόν για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να βοηθήσουμε να προχωρήσει η Ευρώπη, αυτή η απλή Ευρώπη που όλοι θέλουμε άλλο κοινό σημείο και είναι σημαντικό αυτό για τον τύπο και για τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή μέσω του ίντερνετ. Όταν λέμε ότι θέλουμε αυξημένο ρόλο του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι για να δείξουμε ότι να υπάρχουμε και έχουμε περισσότερες εξουσίες. Κάθε άλλο, αν είμαστε σοβαροί, στον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών και πρέπει να είμαστε, αν είμαστε σοβαροί σε θέματα ελέγχου ανισομεριών που δημιουργούνται και αφορούν σημαντικούς τομείς όπως η μισθή, το συζύγιο πληρωμών, οι συντάξεις, τότε χρειάζεται περισσότερη δημοκρατία. Μέχρι στιγμής ε, τα θέματα λυνόντουσαν με ένα είδος αμοιβαίας αδιαφορίας. Ε, παζαρέματα στο, παζαρέματα στο, ε, στο Συμβούλιο, αλογοπαζαρέματα όπως τα λέμε στα αγγλικά, παζάρια στο Συμβούλιο. Αυτό γινότανε. Αν θέλουμε να σταματήσουν τα παζαρέματα χρειάζεται διαφάνεια, χρειάζεται δημοκρατία και το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί στο σημείο αυτό να βοηθήσει κάπως να προχωρήσει η κατάσταση. Ένα άλλο θέμα στο οποίο χρειάζεται εμβάθυνση είναι πρώτον το πολύ λεπτό θέμα των επενδύσεων, προστασία των επενδύσεων προστασία της οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης στην Ευρωζώνη. Γι' αυτό η λέξη να είμαστε προνοητικοί, prudent στα αγγλικά, με, κάπως με προβληματίζει. Με την κορίνη φαντάζομαι θα βρούμε μια λύση. Εγώ δεν θα ήθελα να δοθεί η αίσθηση στον πολίτη ότι μόνο να είμαστε προνοητικοί αρκεί. Δεν αρκεί να είμαστε προνοητικοί ή να είμαστε συνετοί η δουλειά μας είναι να έχουμε μια συνολικά οικονομική ανάπτυξη για όλους και να αυξηθεί το ειδικό βάρος της Ένωσης. Ναι, να είμαστε συνετοί και λελογισμένοι, αλλά χωρίς να αποθαρρύνουμε τις επενδύσεις. Γιατί τα τελευταία χρόνια χάσαμε απόσταση σε σχέση με άλλες χώρες του κόσμου που προηγούνται. Είπε η Ελίζα μίλησε για την εκπαίδευση και για άλλα θέματα. Ένα δεύτερο θέμα που θα ήθελα προσωπικά να μπει στο πακέτο το κείμενό μου ε, μιλάει μόνο για κυρώσεις. Σας καλώ όμως να το δείτε λίγο από απόσταση. Ποια οικογένεια, ποια επιχείρηση, ποια ανθρώπινη ομάδα έχει σαν κίνητρα μόνο κυρώσεις. Δες, ποιο διπάτε, στέλεχος υπεύθυνο για τους ανθρώπινους πόρους και θα σας πει όχι βέβαια. Γι' αυτό εγώ θέλω να ανοίξω και το θέμα των κινήτρων. Κοινών κινήτρων για να σεβόμαστε την πειθαρχία, σας το είπα πριν, γιατί ο στόχος αυτός παραμένει, αλλά να δοθούν κίνητρα, όχι μόνο ο φόβος τιμωρίας και οι κυρώσεις. Αναφέρθηκαν τα ε, ευρωομόλογα, το Financial Times, η Detroit, ε, συζητιέται σε επίπεδο πρωθυπουργών μέσω των εφημερίδων. Το Ευρωκοινοβούλιο θα ανοίξει τη συζήτηση, να δούμε τι δυνατότητες υπάρχουν. Και το λέω για όλους τις συνδεύσεις, ιδιαίτερα αυτούς που έχουν δισταγμούς και τους κατανοώ ο χώρος αυτός της δημοκρατίας πρέπει επιτέλους να ασχοληθεί με αυτό το επίκαιρο θέμα. Επίσης, κάτι άλλο. Όταν καταθέσαμε την έκθεση γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου, δεν ξέραμε τι θα έκανε το Συμβούλιο. Τέλος Σεπτεμβρίου η Κομισιόν είπε ότι ήθελε να αλλάξει τα της οικονομικής διακυβέρνησης με σταθερή συνθήκη. Μετά περάσαμε σε φάση μεταρρύθμισης της συνθήκης. Τα πράγματα κινούνται πολύ γρήγορα. Εγώ δεν είμαι ο φύλακα, ο θεματοφύλακας τη αλήθεια ο μοναδικός, απλώς το επισημαίνω. Για να ενισχυθεί λοιπόν η οικονομική πειθαρχία και έχουν γίνει και σημαντικές ακροάσεις στην Επιτροπή για την κρίση κλπ. Είχαμε άλλη μία στην δική μας Επιτροπή το θέμα των ευρωομολόγων σε σχέση πάντα με την οικονομική πειθάρχηση, το θα είναι blue bonds, red bonds, δεν ξέρω τι θα είναι, πάση περιπτώσει να συζητηθούν όλες οι δυνατότητες προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενο το οποίο είναι αυτό που είναι αυτή τη στιγμή. Άλλο θέμα, δύο θέματα μάλλον που τα θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά προσωπικά. Πρώτον, να δοθεί στην Ένωση και ιδιαίτερα στην Ευρωζώνη μια παγκόσμια διάσταση. Είχαμε ένα πολύ θετικό γεγονός τι τελευταίε εβδομάδε. Η έκδοση των πρώτων ομολόγων EFSF. Δηλαδή ξέρουμε ότι σε αντίθεση με άλλε. Ε, τρελές εισαγωγές του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου η Ευρώπη για τους ξένους επενδυτές κρατάει ακόμα τον βαθμό έλξης, σημαντικό βαθμό έλξης. Αυτό θα μας επιτρέψει να έχουμε χρήματα με λογικά επιτόκια στο διεθνές επίπεδο. Έτσι ώστε το ευρώ να παίξει το ρόλο τον οποίο είχε κλειθεί να παίξει από την αρχή, δηλαδή ένα ρόλο παγκοσμίου νομίσματος. Και το δεύτερο, να επιτραπεί στην τράπεζα, στην κεντρική τράπεζα, που κάτω από δύσκολες συνθήκες πήρε θαραλέες, αμφιλεγόμενες αποφάσεις, ο καθένας ε, μπορεί να έχει τη γνώμη του πάνω σε αυτό, δεν είναι μαυρό πράγματα, αλλά αυτό που έγινε πέρσι ήταν χρήσιμο μέσα στα πλαίσια μιας έντονης κρίσης, αλλά μακροπρόθεσμα πρέπει να έχουμε ένα εργαλείο που να ε, μην ε, επιτρέψει στην κεντρική τράπεζα να γίνει μια bad bank, ε, κακής ποιότητας τράπεζας, τράπεζα η Κομισιόν για δικούς τη λόγους διαχώρισε τα θέματα στρατηγική 2020 και οικονομική διακυβέρνηση ε, ανάκαμψη της εσωτερικής αγοράς. Κατά τη γνώμη όλα αυτά είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο και αυτό το συνολικό όραμα θα πρέπει να το έχουμε συνεχώς κατά νου. Και πιστεύω ότι όλοι μας, όπως το είπαν οι συνάδελφοι ήδη, είμαστε στη διάθεση, στη διάθεσή σας έτοιμοι να ακούσουμε οτιδήποτε από την Ουγγρική Προεδρία, όπω είπε, να με υποστηρίξει θέση του Κοινοβουλίου. Το χρονοδιάγραμμα είναι να κλείσουμε τον Ιούνιο. Πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Δεν το λέω αυτό για να μην τηρηθεί, αλλά χρειάζεται σοβαρή προσπάθεια σύγκληση μεταξύ των ομάδων. Στι τροπολογίε, στι συζητήσει που θα γίνουν από εδώ και μπρο μέχρι τον Ιούνιο, διαφορετικά θα έχουμε δυσκολίε. Η Task Force κινείται ήδη με το δικό τη ρυθμό και όπως είπε ο Ούγκο, το Συμβούλιο δεν λαμβάνει και πολύ σοβαρά υπόψη, δυστυχώς, αυτό που κάνουμε την έκθεση Μπέρενς, με την έκθεση Φεγιό κλπ. Ευχαριστώ και πάλι όλους σας. Ε, ε, ευχαριστούμε. Ο Κάρλ και μετά η Βίκη. Οι σκιώδε που θέλουν να μιλήσουν, σα παρακαλώ να σκόσετε το χέρι να σημειώσετε, γιατί έχω ένα μεγάλο κατάλογο εδώ. Φίλιψ έγραψα. Σημειώνω σημειώνω. Κάρολα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι στον πιο σύντομο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία μέχρι στιγμής και τη γραμματεία και ευχαριστώ ιδιαίτερα την Καρίν για όλες τις συναντήσεις ε, κάτω που ήταν πάρα πολύ σημαντικό σε γενικές γραμμές νομίζω πως πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το πόσο σημαντικό είναι αυτό το πακέτο και για την τωρινή κρίση. Παρά το, το πακέτο δεν θα λύσει την κρίση γιατί αφορά περισσότερο το μέλλον, νομίζω πως είναι σημαντικό να αντιληφθούμε πόσο ουσιαστικό είναι για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο ευρώ και το κοινό νομισμά και μεταξύ των ανθρώπων και βέβαια στις αγορές. Οπότε χαίρομαι που εργαζόμαστε σε αυτό το πακέτο και με φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα. Όσον αφορά την εκθεσή μου που σχετίζεται βεβαίω στενά με την έκθεση της κυρίας Φερέιρα που παρουσιάστηκε ήδη έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον νέο μέρος κάτι το δύσκολο από μακροοικονομική σκοπιάς και εγώ θέλω προσωπικά να επιτύχουμε και είμαι σίγουρος πως το περασμένο έτος έπαιξε πόσο σημαντικό ε, μπορεί να είναι, πόσο σημαντική μπορεί να είναι η Ένωση όσον αφορά τη μακροοικονομική εποπτεία. Ταυτόχρονα εφόσον βεβαίως πάμε σε νέες ανεξαρεύνητες περιοχές πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε με, τις, με την παρακολούθηση και τις πιθανές κυρώσεις έτσι ώστε να θεωρούνται δίκαιες και βέβαιως αποτελεσματικές. Εδώ πέρα είμαι σίγουρος πως ήδη σε αυτά τα οποία έχουμε κάνει οι συγητές έχουμε βελτίωσει κατά πολύ το πακέτο και μπορούμε να κάνουμε ακόμα πολλά πράγματα και είμαι σίγουρος πως οι συναδελφοί που είναι εδώ πέρα και άλλοι θα κάνουν το μακροοικονομικό κομμάτι ακόμη πιο λειτουργικό για το μέλλον, γιατί παρά το ότι ίσως είναι κάπως επίμαχο με μακροοικονομική επιτήρηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, νομίζω πως είναι σημαντικό για όσους ε, είναι επικριτικοί να σκεφτούν ποια είναι η εναλλακτική λύση που είναι να μην το κάνουμε και είναι βεβαίω κάτι πολύ χειρότερο. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο καλύτερα μπορούμε την κατάσταση και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα αξιόπιστο που θα λειτουργεί. Όπω είπα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά με την κυρία Φερέιρα και σχετίζεται η έκθεσή τη με τη δική μα και προσπαθήσαμε εδώ πέρα να έχουμε μια προσέγγιση με την οποία υπογραμμίζουμε την αναγκαιότητα να μπορέσουμε να πείσουμε τα κράτη-μέλη εκείνα μακροοικονομικές ανισορροπίες να θελήσουν τα ίδια να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανισορροπίες πριν ε, γίνει ένα πρόβλημα το οποίο θα διαχειριστεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εδώ λοιπόν νομίζω πως έχουμε επιτύχει και στο να ξεκαθαρίσουμε το ότι δεν προσπαθούμε να τιμωρήσουμε χώρες με προβλήματα, αντιθέτως όπως είπα προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα με το οποίο οι χώρες θα ενθαρρύνονται να κάνουν αλλαγές και ε, η μη, συμμόρφ, η μη λήψη διορθωτικών μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε κυρώσεις, γιατί είχαμε πάρα πολλές παρεξηγήσεις στα ΜΜΕ και στους διαδρόμους εδώ του Κοινοβουλίου. Μετά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι κάπως πιο αυτόματο από αυτό το οποίο επεξεργάζεται το Συμβούλιο και νομίζω πως αν πάμε πίσω το 2005 όταν αναθεωρήθηκε το Συμβούλιο Σταθερότητας και Ανάπτυξη λόγω κάποιων προβλημάτων, νομίζω πως αυτό αποδεικνύει πως χρειαζόμαστε ένα αρκετά αυτόματο σύστημα. Δηλαδή όταν έχουμε μια προφανή περίπτωση να λαμβάνετε δράση και να μην έχουμε πολιτικά παζάρια που οδηγούν σε αλλαγή ή μη χρησιμοποίηση του συστήματος. Προσωπικά θεωρώ πως είναι σημαντικό τα πιθανά πρόστιμα για μη συμμόρφωση να είναι αρκετά σκληρά. Ε, δηλαδή σημαίνει αυτό ότι προτείνω να έχουν μια κλίμακα, να είναι κλίμακοτά αυτά τα πρόστιμα και νομίζω είχαμε ευρεία συνένεση πως όταν μιλάμε για χώρες που παραποιούν στατιστικά στοιχεία ή έχουμε ξεκάθαρες περιπτώσεις απάτης να έχουμε σκληρότερες κυρώσεις 0,5% ε, του ΑΕΠ ταυτόχρονα προσπαθήσαμε να βρούμε έναν τρόπο με τον οποίο θα έχουμε κάποιο πλαφόν στα πρόστιμα γιατί δεν μπορούμε να έχουμε τεράστια πρόστιμα κάτι το οποίο θα έχει φιλοκυκλικό αποτέλεσμα γιατί εν λόγω χώρα. Και τέλος, όπως είπε και η κυρία Φέριο, πρέπει να δούμε το πού θα πηγαίνουν ε, πιθανώς αυτά τα κονδύλια. Το να διανέμονται δηλαδή στις πλουσιότερες χώρες δεν είναι τόσο έξυπνο, οπότε θα μπορούσαν τα κονδύλια να πάνε στο μηχανισμό κρίσης. Στο ταμείο αυτή τη στιγμή δημοσιονομικής σταθερότητας είναι μια καλύτερη λύση κατά την άποψή μου. Οπότε σε γενικές γραμμές νομίζω πως κάνουν αρκετά καλή δουλειά εδώ πέρα και αναμένω τη συζήτηση με τους συναδέλφους, τροπολογίες, διαπραγματεύσεις. Ήδη οι σκιοδησηγητές είναι πολύ δραστήριοι και είμαι σίγουρο ότι θα βρεθεί κάποια συνένεση. Κατά την άποψή μου το σημαντικότερο είναι να έχουμε ευρεία συνένεση στο Κοινοβούλιο, μόνο έτσι θα είμαστε ίσχυροι για να διαπραγματευτούμε με το Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίκη. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη γιατί δεν θέλω εγώ να μιλάω χωρίς σταματημό στους ε, σκιοδησίτες και νομίζω πως πρέπει να γίνει μια δημόσια συζήτηση για τα ζητήματα που φύγονται εδώ πέρα. Οπότε αν δεν έχουμε χρόνο πρέπει να βρεθεί χρόνος κάποια στιγμή. Η έκθεση την οποία εξετάζω είναι μια πρόταση για τις απαιτήσει που εφαρμόζονται στα δύο δημοσιονομικά πλαίσια των κρατών μελών από τις προδιαγραφές λογιστικές μέχρι την ε, διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Βεβαίως και αυτό ε, σημαίνει πως ο σχεδιασμός των προπολογισμών επηρεάζει και το περιεχόμενό τους και πιο αυστηρές διαδικασίες σε εθνικό επίπεδο σημαίνει πως συμμορφωνόμαστε περισσότερο με το σύμφωνο σταθερότητας ε, και άρα όπως είπε και η Σόφνα έχουμε μια πιο βιώσιμη αντιμετώπιση των δημοσίων οικονομικών. Η έκθεση αυτή δεν είναι συναπόφαση, αλλά συνεργάστηκα στενά με τους συζητητές συναδελφού για να διασφαλίσουμε πως κάποιε από τι προτάσεις μου ε, αναφέρονται και αλλού. Όπως ε, βεβαίω είναι αναμενόμενο, άκουσα τους ε, υπόλοιπου συζητητές από την Ευρωζώνη για, για τα σημεία στα οποία θα ήθελα να πάμε ακόμη παραπέρα. Βεβαίως, το θέμα εδώ πέρα είναι η διαφάνεια. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε την ευαισθησία αυτού του θέματος. Οι εθνικοί προπολογισμοί πάντα ήταν αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κυβερνήσεων και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια χρυσή τομή μεταξύ των ορθών πρακτικών και του σεβασμού τη εθνική κυριαρχία στου προπολογισμού. κάτι το οποίο ψηφίσαμε όλοι όταν ψηφίσαμε την ε, έκθεση Και βεβαίως ε, σεβόμαστε τις εθνικές δεσμεύσεις πάνω και πέρα από το ευρωπαϊκό επίπεδο. Οπότε τα πέντε βασικά χαρακτηριστικά αφορά την ε, διαφάνεια και του χρέους και των διαθέσιμων μετρητών και των επισφαλιών, ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει κανείς, το ποιες υποθέσεις γίνονται, η μεθοδολογία και πώς γίνονται οι προβλέψεις. Δεύτερον βεβαίως είναι λογιστικά πρότυπα, το τρίτο είναι ανεξάρτητα δημοσιονομικά όργανα με ισχυρή εποπτεία να φροντίσουμε βεβαίως ε, να είναι προσαρμοσμένοι στην κάθε χώρα, καθώς οι χώρες εκείνες οι οποίες έχουν εθνικούς δημοσιονομικούς κανόνες ε, προσαρμόζονται καλύτερα στο σύμφωνο σταθερότητα και πρέπει εδώ πέρα να σημειώσουμε πως διαφορετικές χώρες έχουν διαφορετικές υποχρεώσεις σύμφωνα με το σύμφωνο αυτό. Το τέταρτον βεβαίως αφορά την ε, ανεξάρτητη εποπτεία στην οποία θα επανέλθω και τέλος έχω ένα κομμάτι για την διαφάνεια. Δηλαδή, αν ζητάμε από τα κράτη-μέλη να έχουν περισσότερη διαφάνεια στο πώς συντάσσουν τον προπολογισμό τους και ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να μπει στην ίδια διαδικασία λόγω της αλληλεξάρτησης των προϋπολογισμών κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε το ίδιο επίπεδο διαφάνειας θα ήταν κάτι το θετικό. Πρέπει να συζητήσουμε επίσης τις προβλέψεις και το συγκεκριμένο ρόλο των προβλέψεων της Κομισιόν. Και πάλι εδώ πέρα η διαφάνεια είναι κλειδί. Δεν πρέπει να γίνεται τίποτα πίσω από κλειστέ πόρτες. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στη μεθοδολογία και στι υποθέσει πίσω από έναν προπολογισμό που θα μπορεί να εξετάζει η Κομισιόν και να κάνει τι δικέ τη προβλέψει για να παρουσιάζει στάσει στα κράτη-μέλη, αλλά τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μπορούν να κάνουν τι δικέ προβλέψει εντό ενό πλαισίου, ακούγοντα την Κομισιόν και του υπολείψεις. Και νομίζω πως ε, καμιά φορά η απόκληση απόψεων ε, μπορεί να είναι κάτι το υγιές. Δεν ε, είναι μια ακριβής επιστήμη αυτή εδώ πέρα, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα έχουν τα κρατημένη λόγο για το τι συμβαίνει. Καθώς βλέπουμε πως εάν θα πρέπει εάν ή προβλέψει των κρατών μελών συνεχώ είναι χειρότερε από αυτέ τι Κομισιόν, θα πρέπει να μπορούν να ε, συμμορφώνονται με αυτέ τι Κομισιόν. Επίση, θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι βέλτιστε πρακτικέ εντό Ένωση ε, Ολλανδία, Σουηδία, Αυστρία και άλλοι. Και πρόσφατα στο Ηνωμένο Βασίλειο εγκρίθηκε ένα ανεξάρτητο φορέα με ευθύνη για τον προπολογισμό. Και έχει αποδειχθεί, υπάρχουν στοιχεία για το ότι τέτοιοι ανεξάρτητοι φορείς μπορούν να έχουν επίπτωση στην δημοσιονομική πειθαρχία. Οπότε εμείς ζητάμε να είναι υποχρεωτικό κάτι τέτοιο εντός της Ευρωζώνης και θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις Συμβουλίου εδώ πέρα. Επίσης, θα πρέπει να σημειώσουμε πως πολλά κρατημέλη ήδη συμμορφώνονται πλήρως με τις περισσότερες συστάσεις στον τομέα αυτών και η Κομισιόν δεν συνιστά καινούρια νομοθεσία, αλλά ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τις δικές τους διαδικασίες. Συμφωνώ με αυτό, αλλά οι συνάδελφοι από την Ευρωζώνη ζήτησαν μια ρήτρα που θα λέει πως θα πρέπει να εισαχθεί ειδική νομοθεσία για την οδηγία εντός της Ευρωζώνης. Τέλος, σύντομα, για τα άλλα σχόλια που ακούστηκαν, η πρόταση του Μάριου Μόντι για κονδύλια που πάνε για μακροχρόνιες επενδύσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από το υπόλοιπο χρέος. Καλή πρόταση, αλλά ποιο ακριβώς είναι το όριο, ποια έργα εμπίπτουν και ποια όχι. Επίσης η εμπειρία που έχουμε είναι πως όταν διαχωρίζουμε τα έσοδα από τις ε, υπόλοιπες επενδύσεις ε, αρχίζουμε ήδη να μπλέκουμε τους εθνικούς λογαριασμούς. Σύμφωνο λοιπόν με την Κορίν πως έχει καλυφθεί. Επίσης για τις ανισορροπίες πρέπει να είναι η ίδια αντιμετώπιση εντός και εκτός της Ευρωζώνης. Εδώ πέρα νομίζω πως ε, μειώνουμε τη σημασία των συνταγματικών ισοτιμιών στην οικονομική πολιτική και δεν συμφωνώ. Και τρίτον, κάτι το οποίο προέκυψε, είναι η πρόταση για να δοθούν περαιτέρω ε, εξουσίες σε έκτακτες ε, περιπτώσεις στην Κομισιόν. Ε, ανησυχώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι κάτι το πολύ ευαίσθητο στο ήδη υπάρχουν πακέτο και θα είναι ακόμη πιο ευαίσθητο στον τομέα του περιβολισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα προχωρούμε στη γενική συζήτηση. Τουλάχιστον εννέα σκιώδεις συζητητές θέλουν να λάβουν το λόγο. Υπάρχουν κάποιοι που είναι σκιώδεις σε πολλές εκθέσεις και όχι μόνο σε μία και άλλους οκτώ ομιλητές και έχουμε λιγότερο από μια ώρα στη διάθεσή μας. Επομένως θα μείνουμε από χρόνο σίγουρα αν θέλετε να πείτε ο καθένας όλα αυτά που θέλετε να πείτε. Θα πρέπει να βρούμε λοιπόν κάποιο άλλο χρόνο για να καλύψουμε τα υπόλοιπα θέματα που δεν θα προλάβουμε να τα πούμε. Ο Φίλιπ, ο οποίος είναι κατ' επανάληψη εισηγητή, είναι πολλαπλό εισηγητή, αλλά πρέπει να σκεφτεί και του άλλου οι οποίοι έχουν λάβουν το λόγο. Ναι, το κατάλαβα, λέει ο Φιλίπ. Απλώ θέλω να συμμεριστώ την κοινή σα άποψη ότι ο στόχο είναι η σύγκληση και είναι εργαλείο η μακροοικονομική εποπτεία. Χωρί τη σύγκληση δεν έχουμε πραγματική οικονομική ε, ένωση, οπότε θα αρχίσει να καταραίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε κάτι τέτοιο, γι' αυτό εμεί θέλουμε να ενισχύσουμε την οικονομική διακυβέρνηση και υποπτία. Αυτό σημαίνει κοινοί κανόνε, ε, κοινά εργαλεία κτλ. Οι έξι αυτέ εκθέσει έχουν αναφέρει πάρα πολλά πράγματα και τα είπαν οι Θα μείνω μονάχα σε έξι σημεία όπου υπάρχουν μείζωνα θέματα. Καταρχήν, η τροχιά σύγκληση. Σύγκληση, το ανέφερε και ο Ούντο. Εγώ σκέφτομαι την ε, έννοια του ενός εικοστού μείωση του χρέους το χρόνο. Για ορισμένε περιπτώσεις μπορεί αυτό να είναι πολύ αυστηρό, σε άλλες περιπτώσεις να είναι πολύ χαλαρό. Η Ελλάδα, παραδείγματος χάρη, για να μπορέσει να το κάνει αυτό, χρειάζεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα του ΑΕΠ 10%. Αυτό είναι αδύνατο, δεν μπορεί να γίνει, το ξέρετε όλοι. Ένα δεύτερο σημείο. Αν δούμε την σημερινή κατάσταση περίπου 20 κράτη-μέλη θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν μια διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος ή υπερβολικής ανισομέρειας και αν όλα αυτά τα κράτη περάσουν σε λιτότητα αυτό διπλασιάζει το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα το οποίο σημαίνει ότι προχωρούμε ακόμα πιο γρήγορα σε μια ύφεση ή σε αρνητική ανάπτυξη, αν θέλετε να μιλάμε για ανάπτυξη, κάτι το οποίο θα πλήξει ακόμα περισσότερο την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Διαβάστε τον οικονομικό τύπο και θα το καταλάβετε. Δεύτερο σημείο, οικονομικές, μακροοικονομικές ανισομέρειες. Εδώ θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι αν δείτε την περίπτωση της Ιρλανδίας και της Ισπανίας, οι περιπτώσεις αυτές δεν είχαν να κάνουν τίποτα με λανθασμένες χειρισμούς Τη κυβέρνηση. Μόνο με τον ιδιωτικό τομέα είχαν να κάνουν και δεν είναι σοσιαλιστική η κοινωνία μα και η οικονομία μα. Επομένω, είναι περιορισμένη η δυνατότητα τη κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τον ιδιωτικό τομέα και τι λαθροχειρίες του. Υπάρχει αυτή η εξουσία, αλλά είναι περιορισμένη. Το να τιμωρούμε κυβερνήσει για κάτι το οποίο δεν ελέγχουν είναι κάτι το οποίο είναι λαθασμένο για μένα. Στην περίπτωση τώρα των φυσαλίδων που, δημιουργήθηκαν και που δημιουργούσαν αυτά τα προβλήματα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει μεγαλύτερη δυνατότητα να τις ελέγξει από ό,τι τα κράτη-μέλη. Επίσης, λέμε ότι πρέπει να είναι υπερκυκλική αυτή είναι υπερκυκλική αυτή η διαδικασία που προτείνουμε και δεν δίνουμε καθόλου κίνητρα. Τα ευρωμόλογα μπορούν να είναι ένα είδος κινήτρου, αλλά είμαστε ακόμα πόρο μακριά από αυτή την αντιμετώπιση. Επίσης έχουμε μια ενιαία αντιμετώπιση για όλους και δεν έχουμε αποτρεπτικούς παράγοντες. Πέμπτο σημείο. Το πακέτο αυτό, λόγω της ε, κοινοτική μεθόδου που την υποστηρίζουμε εμείς, θα πρέπει να δώσει περισσότερη εξουσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε τυφλοί στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα πολιτικό σώμα, δεν είναι τεχνοκράτες. Και αυτό καταδεικνύει και η αιτήσια επισκόπηση για την ανάπτυξη που λέει ότι για να ξαναγυρίσουμε σε βιώσιμη οικονομία πρέπει να αναθεωρήσουμε τις ε, αγορές εργασίες και να μειώσουμε τις δημόσιες δαπάνες, τίποτα για επενδύσεις στο μέλλον, τίποτα για σύγκληση, ούτε ακόμα και όταν έχουμε ξεκαθαρίσει τα προβλήματα των οικονομικών μας. Έκτο σημείο και τελευταίο και λουκούμιο αφορά την Γενική Διεύθυνση Μονάχα Οικονομικών. Οι άλλες γενικές διευθύνσεις δεν θα έχουν καμία σχέση. Παραδείγματο χάρη, έχουμε εκθέσει για την αγορά εργασία, αυτό είναι η Γενική Διεύθυνση Απασχόληση πρέπει να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Αλλά το παιχνίδι το καθορίζει η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά στην Κομισιόν. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που έχουμε να κάνουμε και όλο αυτό το πακέτο βασίζεται σε μία υπόθεση ότι επειδή δεν μπορούμε να έχουμε πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση, χρειαζόμαστε κανόνες που θα υποκαταστήσουν αυτή τη διακυβέρνηση. Και αν δεν στέκεται αυτό, για είναι λαθασμένη αυτή η υπόθεση. Αν είναι αδύνατο να υποκαταστήσει κανείς την πραγματική ευρωπαϊκή διακυβέρνηση που τη χρειαζόμαστε για να ευδοκιμήσει η νομισματική ένωση με κανόνες τέτοιου είδους οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν γιατί έχουν αποδείξει στο παρελθόν ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν και εγώ πραγματικά αμφιβάλλω ότι μπορούν να υποκαταστήσουν μια πραγματική οικονομική διακυβέρνηση. Σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν δεν πρέπει να παραιτηθούμε από την ιδέα αυτή ότι ίσως θα πρέπει να προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά και να κάνουμε αυτό το οποίο ο Τρισέ ανέφερε επιφυλακτικά ως μια ομοσπονδία προπολογισμού, επί του προπολογισμού. Θέλω, εν πάση περιπτώσει, κλείνοντα να ευχαριστήσω του συζητητέ που δουλέψαν με ένα τρόπο ο οποίο ήταν πάρα πολύ περιεκτικό για μία φορά η ομάδα των εισηγητών έχει μεγαλύτερο αριθμό γυναικών παρά ανδρών, αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτικέ αποχρώσεις και διαφορέ μεταξύ μα, αλλά πρέπει να εργαστούμε όλοι από κοινού και επικοδομητικά για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία λειτουργική και ισορροπημένη λύση. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ο κατάλογο των ομιλητών, για να ξέρετε μονάχα ότι δεν έχω ξεχάσει κανένα. Κασία Μαγκάγιο, Ντόφιν, Χουντής και Κάριντς και μετά θα περάσουμε στους ομιλητές οι οποίοι δεν είναι σκιώδεις συζήτητες και θα μιλήσω εγώ, ο Κλίντς, Γκούναρ Χόκμαρκ, Περβάνος Περές, Λούνινγκ, Σφέν Γκίγκολτ και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος άλλος. Εντάξει, ο Ντέρκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνήθως και γενικά υποστηρίζω το πακέτο αυτό για την οικονομική διακυβέρνηση. Πρέπει να το έχουμε σε σχέση πάντα με το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη. Αν δούμε όμως την έκθεση τη κυρίας Γκουλάρτ, την ενίσχυση τη δημοσιονομική υποπτίας, υπάρχει ένα που ε, πάρα πάρα πολύ σημαντικό φαίνεται είναι το θέμα, το θέμα των ευρωομολόγων. Εκτό τόπου θα έλεγα στην περίπτωση αυτή του Ευρωμόργου. Δηλαδή, γράφω μια έκθεση για πρόταση της Κομισιόν και μέσα στην έκθεση βάζουμε μια άλλη έκθεση για ένα άλλο θέμα. Ευρωμόλογα. Άλλο ευρωμόλογο, άλλο ευρωχρέο. Πώ είναι δυνατόν να έχουμε υποπτία τον προπολογισμό, δημιουργώντα επιπλέον χρέο. Αυτέ οι παράγραφοι λοιπόν όπως επίσης και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, γράφηκαν κατά κάποιο τρόπο με βάση το πνεύμα Σπινέλη. Εγώ πηγαίνω όταν η Επιτροπή Σπινέλη οργανώνει διάφορε εκδηλώσει και αναγνωρίζω γι' αυτό το λόγο τη γλώσσα. Αυτή είναι η γλώσσα, ε, η χαρακτηριστική τη ομάδα αυτή. Λάθο δρόμο έχουμε πάρει όμω, αν θέλουμε να το βάλουμε αυτό μέσα στο πακέτο. Γιατί θα θέσει σε κίνδυνο το πακέτο. Αν δεν συμφωνεί η Γερμανία, δεν θα έχουμε ευρωομόλογα. Άκουσαμε τη μαγική ε, λέξη από τον κύριο Κίνκελ. Το κόμμα του σε λίγο θα έχει πολύ δύσκολες εκλογές, σε ένα-δυο μήνες. Αν είστε υπέρ των ευρωμολόγων, τι θα γίνει. Και για την κυρία Βότμαν Κόλ, το ίδιο πράγμα. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο πρόβλημα. Μερικοί φύγανε ήδη, φύγανε ήδη από την αίθουσα. Τα ευρωομόλογα θα βάλουν σε κίνδυνο το πακέτο. Παρακαλώ λοιπόν από τους συγητές και συγγήτρες να ξαναγράψουν την έκθεση. Αυτό το σημείο για τα ευρωομόλογα και το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο να φύγει. Ας κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας. Ναι, μην δημιουργήσουμε τέτοιου κινδύνου. Μα θυμίζει τον προπολογισμό του 2011. Ο καθένα έκανε προτάσει και προτάσει και τελικά όλοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν όπω ο Μεξικανικό στρατό. Το ίδιο πράγμα θα συμβεί και εδώ. Μην αναλάβουμε τέτοιο κίνδυνο. Όσον αφορά τα ευρωομόλογα, το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, Κατά τη γνώμη μου αυτό, αν υπάρχει μέσα στο πακέτο, εγώ δεν συμφωνώ καθόλου. Πρόεδρος, ο Ούντο. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Κομισιόν έχει αυτή τη στιγμή με το πακέτο αυτό μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ή είχε μια μεγάλη ευκαιρία. Γιατί σε όλους τους ευρωπαϊκούς φορείς και στο ίδιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν σαφές ότι μετά από την παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, την κρίση πραγματικής οικονομίας και την κρίση του χρέους, ότι υπήρχε η ανάγκη να ξεπεράσουμε αυτές τις κρίσεις και εφόσον είχαμε ήδη αναλάβει το ιδιωτικό χρέος των πολλών τραπεζών, ήμασταν έτοιμοι να προχωρήσουμε προς μια κοινή δράση, μια κοινή διαδικασία για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. και να μπορέσουμε να έχουμε ένα τρόπο διακυβέρνηση στον οικονομικό χώρο που να είναι επωφελής. Χάσαμε αυτή την ευκαιρία. Το πακέτο αυτό το οποίο έχουμε ενώπιόν μας δεν ουσιαστικά αντιμετωπίζει την ε, κρίση και τις συνέπειές της. Είναι σαν να το γράφει κάποιος από την Κομισιόν, ο οποίος θα το έγραφε είτε υπήρχε κρίση είτε όχι. Δυστυχώς είναι έτσι. Δυστυχώς έχουμε χάσει την ευκαιρία θα πρέπει να βελτιώσουμε λοιπόν αυτό το πακέτο, αλλιώς δεν θα σημαίνει καμία πρόοδο στην ε, οικονομική διακυβέρνηση της Ευρώπης, ό,τι αφορά τα σημεία που υπάρχουν πραγματικές ελλείψεις. Δεν έχει καθόλου ιδέες για το πώς μπορούμε να βγούμε και να ξαναπεράσουμε στην ανάκαμψη σε μια τέτοια κρίση. Δεν υπάρχει το στοιχείο της ανάκαμψης. Το στοιχείο της ανάκαμψης. Όλες τις προτάσεις κομισιών το παραλείπουν αυτό το στοιχείο η κυρία Γκουλάρ, θα πρέπει να ξέρει ότι δεν είναι μονάχα το θέμα του να διατηρήσουμε τις επενδύσεις. Υπάρχουν πολλές χώρες στις οποίες θα πρέπει να υπάρξουν πολύ περισσότερες επενδύσεις για να μπορούμε να δημιουργήσουμε δυνατότητες ανάπτυξης στο μέλλον. Και η κυρία Βόρτμαν Κόλ νομίζω ότι έχει ένα διαρθρωτικό σφάλμα στην επιχειρηματολογία της. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επενδύσεις, αλλά αυτό δεν πρέπει να αναφέρεται μονάχα μαζί με τις διαρθρωτικές αλλαγές. Δεν μπορούμε να έχουμε λοιπόν μόνο για τις ε, μεταρρυθμίσεις. Το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε επενδύσεις οι οποίες είναι λογικές, ώστε κάποια στιγμή να βγούμε από αυτό το βουνό του χρέους που έχουμε, χωρίς να κάνουμε σμπαραλιά την οικονομία μας. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσει η Επιτροπή μας. Αν δεν υπάρξει καμία μεγάλη πλειοψηφία στην Επιτροπή μας που να ακολουθήσει μια αντίθετη άποψη, δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε από την άποψη της ε, Κομισιόν. Υπάρχει το ερώτημα πώς πρέπει να λειτουργεί κανείς σε ένα οικονομικό κύκλο. Καταρχήν θα πρέπει να καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει ο οικονομικός κύκλος. Δεν μπορεί να υπάρχει ποτέ ένα πακέτο το οποίο λειτουργεί σε οποιαδήποτε φάση του οικονομικού κύκλου. Πρέπει λοιπόν να συμπεριλάβουμε αυτό το στοιχείο και πρέπει να έχουμε και τη δυνατότητα να είμαστε ευφυείς. Και αυτό δεν σημαίνει αυτόματα μονάχα να αντιμετωπίζουμε και αυτόματα να διακυβέρνουμε. Δεν υπάρχει καμιά γλώσσα όπου η ευφυΐα συμβαδίζει ή συμπίπτει με τον αυτοματισμό. Ο αυτοματισμός είναι η συνεχής μηχανιστική, η μηχανιστική αντίδραση μιας, μηχα, μηχανής σε ίδιες συνθήκες. Ενώ η ευφυΐα των ανθρώπων είναι αυτή η οποία μας επιτρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μεταβαλλόμενες και διαφορετικές συνθήκες. Και αυτό μου λείπει στις εκθέσεις των ε, εισηγητών. Επίσης και η αρχή του να μπορούμε να επιβάλλουμε φόρους για να μπορούμε να βγούμε από την ε, κρίση και από την υπερχρέωση. Αυτό είναι κάτι το οποίο λείπει στην πρόταση της Κομισιόν η αυτόματη ε, οι αυτόματοι σταθεροποιητέ στην ευρωπαϊκή οικονομία θα έπρεπε να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Αλλά το γεγονός ότι εμείς περικόπτουμε όλες τις κοινωνικές παροχές είναι ο λαθασμένος τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα της κρίσης. Οι επενδύσει θα πρέπει να έχουν σαν στόχο να λειτουργήσει η Ευρωζώνη. Υπήρξαν αυτέ οι αναφορές για τη γερμανική κατάσταση αλλά και πάλι εδώ πρέπει να πω ότι δεν πρέπει από κάθε, από την τελευταία δημοτική εκλογή να παίζεται το μέλλον της Ευρώπης επειδή και μόνο η Γερμανία είναι το μεγαλύτερο κράτος μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει και η ίδια η Γερμανία να λειτουργεί με βάση ευρωπαϊκά κριτήρια και όχι μονάχα η κυβέρνηση να σκέφτεται αν θα χάσει μια περιφερειακή ή τοπική εκλογή την επόμενη Κυριακή. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις για το τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να γίνει σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλουμε, αλλά δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να είμαστε ενωμένοι σε αυτήν την ε, θέση η οποία θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να έχουμε κοινέ τροπολογίε οι οποίε θα είναι επικοδομητικέ και βελτιωτικέ και σα ευχαριστώ. Ο Ζωζέ. Ο Χωσέ, μάλλον. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι ιδιαίτερα λακωνικό στα σχόλιά μου. Το πρώτο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε για θέματα οικονομίας, αλλά κυρίως και για θέματα πολιτικής. Αρκεί να δει κανείς τι έγινε στις αγορές όταν ανακοινώθηκε ο προσωρινός μηχανισμός του και το γεγονός ότι θα διευρυνθεί και θα ευκαμπτοποιήσει τη δράση του. Είδατε ότι μειωθήκαν τα στοιχήματα κατά του ευρώ και κερδοσκοπία. Όλοι μας προσπαθούμε πάντα να <laughs> να κάνουμε ιονοσκοπία με τις δηλώσεις των Γερμανών ηγετών, όπως κάναν οι Ρωμαίοι με τις πάλες των αρνιών. Αλλά έχουμε ένα σύνολο πραγμάτων που έχουν ε, λάβει χώρα από τότε που ξεκίνησε το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση και πρέπει να τα συμπεριλάβουμε, αλλιώ θα είναι τελείως ξεπερασμένο αυτό το οποίο θα πούμε. Προφανώς πρέπει να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό εξ, εξάμεινο, για τα ευρωομόλογα, θα πρέπει να ξέρουμε ποια θα είναι η θέση της Ευρωπαϊκής κεντρική τράπεζας, η οποία ήδη αγοράζει δημόσιο χρέος για να ανακουφίσει τις αγορές. Αλλά αν γίνουν όλα αυτά θα γίνει αυτό το οποίο λένε οι Αμερικανοί μια bad bank, δηλαδή μια τράπεζα η οποία έχει βάλει στο θησαυροφυλάκιό της όλα τα αμφίβολης αξία ε, αξιόγραφα. Επομένως, εγώ είχα πει και το γνωρίζει πολύ καλά η Κορίν, ότι η πολιτική απάντηση των κυβερνήσεων στις συστάσεις που κλείνουν το ευρωπαϊκό εξάμεινο θα έχουν σαν στόχο να έχουν μια διαφοροποιημένη αντιμετώπιση κυρώσεων, εάν υπάρχουν κυρώσεις, και να λάβουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση ενός κράτους και να δουν αν ένα τμήμα του δημοσίου χρέους της μπορεί να καλυφθεί από ευρωομόλογα ή όχι το θέμα του μηχανισμού διάσωσης που είναι το κεντρικό θέμα το οποίο μας απασχολεί αυτή τη στιγμή όταν αναφέρθηκε ότι ο μηχανισμός αυτό θα τεθεί σε εφαρμογή το 2013 και ότι με τον τρόπο αυτό μπορεί να υπάρχει το λεγόμενο haircut ή οι μειώσεις των απαιτήσεων για τους ιδιωτικού ε, ιδιωτικούς δηλαδή ο κίνδυνος να συμβαδίζει με μείωση των απαιτήσεων, όπως γίνεται πάντα, το μεγάλο κέρδος μάλλον με τη μείωση των απαιτήσεων, τότε ο, ελέγχθη ότι ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις θα γίνεται με κατά περίπτωση και ακολουθώντας τα κριτήρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η μόνη περίπτωση λοιπόν που εφαρμόστηκε αυτό το λεγόμενο haircut ήταν το 2004 στην Αργεντινή του Κίσνερ. Αυτό οδήγησε σε χάος οι επενδυτές δεν πήραν πίσω τα λεφτά τους και η εμπειρία αυτή είναι, ήταν αρνητική. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την δυνατότητα των ευρωομολόγων. Ίσως η λέξη ευρωομόλογα δεν είναι ιδιαίτερα ε, πρόσφορη, αλλά τα ευρωαξιόγραφα δεν θα πρέπει να είναι μια διαδικασία για να χαλαρώσουμε την ε, λιτότητα και την πειθαρχία του προπολογισμού, αλλά ίσα ίσα για να την ενισχύσουμε. Καταρχήν θα πρέπει να θεσπίζουμε ένα όριο για το δημόσιο χρέος το οποίο θα είναι μέσα σε πλαίσια εγγύησεως και οτιδήποτε ξεπερνάει αυτό το επίπεδο θα πρέπει να καλύπτεται από, ευρωπαϊκ... από, εθνικές, από εθνικά ομόλογα με υψηλά επιτόκια όπως μπορεί κανείς να περιμένει και επίσης αν διατηρήσουμε την έννοια της χρηστής οικονομικής διακυβέρνησης όπως λέει ο Ναπολεωνικός κώδικας, όπως θα κάνει ένας καλός οικογενειάρχης, αυτό, μια τέτοια καλή διαχείριση θα πρέπει να είναι προϋπόθεση για τις χώρες οι οποίες θα την χάνουν εγγυήσεως από αυτό το μηχανισμό. Επίσης, δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε μόνο το δημόσιο χρέος, αλλά το δημόσιο χρέος το οποίο ξεπερνάει τα όρια τα οποία μας φαίνονται ότι είναι λογικά εύλογα. Δηλαδή ό,τι δεν καλύπτεται σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί θα πρέπει να επεμβαίνουν τα ευρωπαϊκά ομόλογα. Τώρα, η ιδέα του Διεθνούς Νομισματικού, του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, θα πρέπει αυτό το ταμείο να εκδίδει ομόλογα και να διανέμει κονδύλια στα κράτη-μέλη και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να έχουμε μια αντιμετώπιση η οποία αντικαθιστά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι αυτό το οποίο ελέγχει τη διαδικασία και ελέγχει τα ειδικά ομόλογα, όπως προτείνεται από την Κομισιόν, θα έχουμε ουσιαστικά ένα τεράστιο μηχανισμό που θα είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα επενδύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επειδή μιλάμε για πολιτική, πρέπει να τονίσουμε στους πολίτες μας ότι θέλουμε την πειθαρχία, αλλά συγχρόνως θέλουμε να έχουμε και την ανάπτυξη. Η ανάπτυξη με τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι εντυπωσιακή. θα είχαμε, αν είχαμε δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ταμείο αυτού του είδους, θα είχαμε ένα είδος σχεδίου Μάρσελ. Αν είχαμε καταφέρει να έχουμε ευρωομόλογα αυτού του είδους που να πηγαίνουν προς συγκεκριμένα σχέδια, θα είχαμε το αντίστοιχο του σχεδίου Marshall. Γι' αυτό η δική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα σαν ένα σύνολο, ας τα συζητήσουμε σαν ένα πολιτικό θέμα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει αν η έξοδος από την κρίση πρέπει να γίνει μεμονωμένα από κάθε χώρα ή αν θα πρέπει να γίνει με αλληλέγγυο τρόπο και συνολικά. Και αν θέλουμε να έχουμε μονάχα κυρωτικά μέσα ή αν θα έχουμε και κίνητρα θετικά για αυτούς οι οποίοι συμμετέχουν θετικά σε προγράμματα σταθερότητας. Right. Okay. Um, Ωραία. Ο κύριος Ντόρφμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω σύντομα κάποιες σκέψεις για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες. Έχουμε εδώ πέρα βεβαίως ένα νέο μέσο. Ένα μέσο για το οποίο πρέπει να διδαχτούμε από το παρελθόν και αυτό σημαίνει για μένα πως η έλεγχη αυτή ε, κατ' ουσίαν ε, των ε, ισορροπιών είναι αποστολή της εκτελεστικής εξουσίας και άρα της Κομισιόν. Και νομίζω πως έχουμε μια καλή πρόταση εδώ πέρα. Π.χ. το ότι προτείνεται μια αντίστροφη ειδική πλειοψηφία είναι κάτι το οποίο θεωρώ εδώ πέρα σωστό. Αλλά Βεβαίως η δική μας η αποστολή ως ε, συνομοθέτη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να επιτελέσουμε και θεωρώ πως θα πρέπει να έχουμε τουλάχιστον τον ίδιο ρόλο με το Συμβούλιο. Κάτι το οποίο με την πρόταση αυτή δεν διασφαλίζεται και θα πρέπει να ζητήσουμε κάποιες βελτιώσεις ως Κοινοβούλιο. Θεωρώ πως η Κομισιόν πρέπει να έχει την απαραίτητη ευελιξία για τον ορισμό των μακροοικονομικών ε, κριτηρίων και βεβαίως θα πρέπει ε, να έχει την ελευθερία να εγκρίνει εδώ πέρα μέτρα το Κοινοβούλιο είναι η συνυπευθυνότητα την οποία έχει αλλά πρέπει θεωρώ εγώ να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις συνθήκες όσον αφορά αυτούς τους δείκτες. Ε, συμφωνώ λοιπόν πλήρως με τους προλήσεις πως Όσον αφορά τον έλεγχο των μακροοικονομικών ανισορροπιών θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου και το ζήτημα της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας αλλά από την άλλη ε, η ανάπτυξη και οι θέσει εργασία δεν θα πρέπει να είναι δικαιολογία των κρατών μελών για να αυξήσουν ε, και να έχουν τεράστιες τέτοιες ανισορροπίες. Γιατί κοιτώντα την Ευρώπη βλέπουμε πως ε, υπάρχουν, σε χώρες, υπάρχουν στις χώρες εκείνες ε, αρκετά μεγάλη ανάπτυξη και αύξηση των θέσεων εργασίας, οι οποίες όμως στηρίζονται σε μη βιώσιμες πολιτικές, οπότε μετά χάνονται πάλι οι θέσεις εργασίας. Επίσης, ε, όσον αφορά τις κυρώσεις, δεν μπορούν αυτές να είναι να έχουν τη μορφή της ε, τιμωρίας, οπότε θεωρώ πως το κλιμακωτό μοντέλο της Κομισιόν ε, έχει πάρα πολύ καλές ε, προσεγγίσεις όσον αφορά την κατανομή των κυρώσεων. Τέλος, κάποιες σκέψεις για την Eurostat και ή την και βεβαίω την ε, δυνατότητα κάποιων κρατών μελών να τη χρησιμοποιήσουν στον βράδυ νομισματική τους πολιτική νομίζω και τις ε, χώρε βεβαίω εκτός Ευρωζώνης νομίζω πω θα πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε οι έξι εισηγητέ και οι εισηγήτριε δύσκολο το έργο του. Πήρα μέρο και σε μερικέ από τι συνεδριάσει και το ξέρω. Και γίνεται μια προσπάθεια να επιτευχθεί μια κοινή γραμμή στι έξι αυτέ εκθέσει και έχουμε και ένα σφιχτικό χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε. Έχουμε πολλέ επικαλύψει. Με έναν υπέρβαρο μηχανισμό, με ένα σωρό επαναλήψει μερικές παράγραφοι που αναφέρονται στο ίδιο θέμα στις έξι εκθέσεις, καλό θα είναι να πάρουμε την πιο σαφή διατύπωση, την πιο λιτή διατύπωση και να διαλέξουμε αυτή την επιτυχή παράγραφο και να αφήσουμε τις άλλες, τις άλλες εκδοχές εννοώ. Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι νομίζω ότι εδώ δίνουμε έμφαση περισσότερο σε πρόληψη και όχι στην επίλυση της κρίσης. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Βρισκόμαστε στην κρίση μέσα και προσπαθούμε να βρούμε μια διέξοδο. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να μιλάμε αν τα πράγματα πηγαίναν καλά, τι θα κάναμε για να προλάβουμε μια κρίση χωρίς κυρώσεις ή αν υπήρχαν κυρώσεις πώς θα λειτουργούσε σαν κίνητρα, σαν αντικίνητρα. Το θέμα είναι ότι όταν έχουμε μια κρίση Μπορεί να διαπιστώσουμε εκεί τότε ότι είναι πολύ σκληρά αυτά τα, αυτές οι κυρώσεις. Το θέμα είναι ποιες είναι οι κυρώσεις που κρατάνε μια χώρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο σε κατάσταση φόβου. Κυρίως είναι οι αγορές που το δημιουργούν αυτό. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν, έχουμε υπερβολικά σκληρές κυρώσεις και μετά πάμε να τις αποδυναμώσουμε κατά κάποιο τρόπο με διάφορα πολιτικά ή διοικητικά ή άλλα μέτρα, καλύτερο θα είναι ευθύ εξ αρχή να μην είχαμε τέτοιου είδου σκληρέ κυρώσει. Δεύτερο, ο ρόλο των κρατών μελών που είναι εκτό τη Ευρωζώνη. Κατά κάποιο τρόπο έχουμε και του ενδιάμεσου. Αυτοί που είναι μέσα στο, στο, στο σύστημα της ε, διετία του ευρωπαϊκού συστήματος που του επιτρέπει να μπουν κάποια στιγμή στην Ευρωζώνη. Τι γίνεται με τι χώρε αυτέ. Αυτέ οι χώρε θα του αφορά ο μηχανισμός χωρίς κυρώσεις ή όχι. Πρέπει να γίνει και μια αναφορά σε αυτό που λέμε ERM2. Όλες οι χώρες, με εξαίρεση ορισμένες, όλες έχουν δεσμευτεί κάποια στιγμή στο μέλλον να μπουν στο ευρώ. Δεν πρέπει να τους φέρουμε και αυτούς όλους μέσα στην οικογένεια. Να δούμε όμως πιο πριν τι κανόνες θα ισχύσουν για αυτούς. Τρίτο, για να βγούμε την κρίση. Έχουμε τη γνωστή οικονομική εξίσωση που λέει ότι χρειάζεται πρωτογενής Πρωτογενέ πλεόνασμα. Δεύτερον, ο ρυθμός οικονομική ανάπτυξη πρέπει να είναι πιο μεγάλο από τα επιτόκια. Και τέλο η απαλλαγή από το χρέο, η κατάργηση του χρέου, το bailout όπω λένε οι Άγγλοι, πρέπει να ληφθεί και αυτό υπόψη. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Το πρωτογενέ πλεόνασμα αυτή τη στιγμή πάμε να το πετύχουμε με προγράμματα λιτότητα. Τα οποία με τη σειρά του μέχρι στιγμή και οι περισσότερε μελέτε που έχω διαβάσει αυτό μα λένε, χειροτέρεψαν τις ε, οικονομικέ επιδόσει όλων των χωρών. Μπορεί μακροπρόθεσμα να έχουν άλλο αποτέλεσμα. Μέχρι στιγμή η εμπειρία μα δείχνει και οι οικονομολόγοι αυτό μα λένε Ιρλανδία, Ελλάδα και άλλε χώρε δεν θέλουν να μπω σε λεπτομέρειε. το αποτέλεσμα είναι αρνητικό μέχρι στιγμή με τα προγράμματα λιτότητα. Μετά είναι το θέμα των επιτοκίων. Η ανακούφιση όσον αφορά το χρέο και τα ομόλογα και ο μόνιμο μηχανισμό θα βοηθήσουν τα πραγματικά επιτόκια των κυβερνήσεων που δανείζονται να είναι χαμηλά. Να βοηθήσουν κάπως την οικονομική ανάκαμψη. Το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Φυσικά πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Γιατί θα έχουμε την αλλαγή της συνθήκης που μιλάει για έναν μόνιμο μηχανισμό σταθερότητας. Από τα λίγα που έχω κάνει και ξέρω τώρα, το θεωρώ πολύ περιοριστικό. Και πιθανότητα μην ισχύσει για όλα τα μέλη τη Ευρωζώνης, ιδιαίτερα για του μικρού. Εσθονία, Μάλτα, Κύπρο. Μόνο αν δείξουν σαφώ ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται σε κίνδυνο, ο μηχανισμό δεν θα ενεργοποιηθεί. Τι είδου οικογένεια είναι αυτή, όταν τα κράτη-μέλη συμβάλλουν στο μηχανισμό και όταν το χρειάζεται, μόνο να αποδείξθει ότι κινδυνεύει το ευρώ, δεν θα ωφεληθούν από αυτό το μηχανισμό. Θα ήθελα διευκρινήσει γι' αυτό για το ΕΕ και το μηχανισμό. Είναι ανεξάρτητος από τις Κομισιόν, είναι τμήμα της Κομισιόν, θα ασκεί την εποπτεία, θα εκδώσει ευρωμόλογα, θα πάρει μέρος σε κινήσεις μείωσης του χρέους ή ε, διαγραφής του χρέους κλπ. Όλα αυτά αποτελούν κομμάτι της εξίσωσης. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, Ζητήσαμε κάποιες συμβουλέ για την διατύπωση της συνθήκης, για αυτό ακριβώς το οποίο λε, για το τι απειλεί την Ευρωζώνη στο σύνολό τη, γιατί εγώ θεωρώ πω είναι σημαντικό θέμα που πρέπει να, να δούμε. Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζω. Κατόπιν ο κύριος Χουντή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, είμαι ο σκιώδης συγητή εκ μέρου τη ομάδα στις 3 από τις έξι εκθέσεις, τις τρεις τελευταίες κατά τη σημερινή, κατά τη σημερινή παρουσίαση. Με αυτή την έννοια, ό,τι πω δεν έχει καμία σχέση με την προσπάθεια που κάναν οι εισηγητές, φιλότιμοι, την παρακολούθησα από κοντά, αλλά έχουν να κάνουν με τη γενική σύλληψη του θέματος και με το αυτό που ονομάζεται οικονομική διακυβέρνηση. Και να σας πω ότι εκ μέρους της ΓΚΟΕ, το έχουμε ξανακουβεδιάσει, είμαστε ριζικά αντίθετοι. Φοβάμαι ότι μπαίνοντα σε αυτά τα συμπεράσματα της Επιτροπής, υιοθετώντα δηλαδή την άποψη ότι δεν θα έχουμε κρίση, θα μπορέσουμε να προλάβουμε ανισορροπίες, αν κάνουμε πιο αυστηρό το σύμφωνο σταθερότητας και αν αποκαταστήσουμε ένα μηχανισμό μακροοικονομικών ανισορροπιών, πάμε σε λάθος κατεύθυνση. Εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας εν μέρη, αλλά η Επιτροπή της κρίσης έχασε την ευκαιρία να κάνει σωστή διάγνωση των αιτιών της κρίσης. Ενώ ξεκινήσαμε καλά, οι, οι διαπιστώσεις μετά δεν μας βοήθησαν. Αυτή ήταν χαμένη ευκαιρία. Τώρα όμως δεν είναι χαμένη ευκαιρία. Τώρα έχουμε συνευθύνη για το πού θα οδηγήσει η εφαρμογή αυτού του πακέτου. Να είμαι πιο αναλυτικός για να γίνω ίσως και πιο κατανοητός. Με αυτό το πακέτο λοιπόν επιδιώκεται η αυστηροποίηση του πλαισίου άσκησης οικονομικής πολιτικής. Και τι συμβαίνει με αυτή την υπόθεση. Θα χρησιμοποιηθεί αυτό το πακέτο ως μοχλός πίεσης απέναντι στα κράτη να κάνουν βαθιές, βίαιες αλλαγές σε πλευρές της οικονομικής πολιτικής και βεβαίως όλη αυτή την υπόθεση θα την πληρώσουν οι εργαζόμενοι και η πλειοψηφία των κοινωνιών και θα σας πω γιατί. Πρώτος άξονας. Στο όνομα να ελέξουμε τα ελλείμματα και να μην έχουμε τόσα ελλείμματα και χρέος που σημαίνει ένα πιο αυστηρό σύμφωνο σταθερότητας με κυρώσεις θα έχουμε τα αποτελέσματα που είχε και που θέλουμε ενδεχομένω να δούμε το σύμφωνο σταθερότητας. Σε αρκετέ δηλαδή εκθέσει, αρκετοί συνάδελφοι λένε ναι σε αυτό τα ελλείμματα, αλλά να έχουμε και ανάπτυξη να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τη απασχόληση. Από τι αυταπάτε, α το πω έτσι επίοικο, τη στρατηγική τη Λισαβόνα, που σύμφωνο σταθερότητα και πλήρη απασχόληση όπω υπόσχονταν, δεν έχουμε φύγει. Αυστηρό σύμφωνο σταθερότητα και απασχόληση και ανάπτυξη δεν μπορεί να γίνει. Δεύτερη πλευρά αυτού του ζητήματο. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η Κομισιόν και οι εισηγητέ μέσα σε αυτό το πλαίσιο εισηγούνται κυρώσει. Σε αρκετέ περιπτώσει οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτέ οι κυρώσει έχουν φιλοκυκλικό χαρακτήρα. Αντί να αντιμετωπίζουν τι ανισορροπίε, πιθανόν να τι διευρύνουν. Πάμε στο μηχανισμό για τι ανισορροπίε. Εκεί βάζονται πρόβλεψη. Εκεί βάζονται διάφορα στοιχεία πρόγνωση που προβλέπουμε ή που θα έχουμε ανισορροπίε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πολλοί από αυτού του δείχτε όπως ας πούμε το εμπορικό ισοζύγιο, δεν ελέγχεται απόλυτα από τα κράτη και τις κυβερνήσεις. Και ποιο θα είναι τώρα το αποτέλεσμα. Επειδή δεν μπορεί να το ελέξει, θα λέμε κάνε, έχουμε την εμπειρία της Ελλάδας τώρα πια και της Ιρλανδίας, κάνε διαρθρωτικές αλλαγές στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά και ούτω καθεξής. Είναι ο ισχυρισμό που σας είπα που θα καταλήξει αυτός ο μηχανισμός. Με αυτές τις βασικές παρατηρήσεις είναι φανερό ότι είμαστε σε λάθος κατεύθυνση φιλότιμες προσπάθειες με τον ένα ή τον άλλον τρόπο που γίνονται, κάποιες νέες ιδέες, θα σας έλεγα θα μπορούσε κανείς να τις συζητήσει όπως ας πούμε Ευρωπαϊκό Ενιαίο Νομισματικό Ταμείο, θα μπορούσε να το συζητήσει κανείς, αλλά σε ένα διαφορετικό πλαίσιο. Θα μπορούσε να το συζητήσει κανείς όχι σαν αντιγραφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Θα μπορούσε να το συζητήσει κανείς ως ένα ταμείο αλληλεγγύη, όχι ω ένα πλαίσιο που θα το πληρώνει πανάκριβα, όπω γίνεται σήμερα με του μηχανισμού ε, ε, λεγόμενης στήριξης. Και άλλα θα μπορούσα να αναφέρω. Εκεί μέσα τώρα, μέσα από όλο το πακέτο, τι βγαίνει, που, δεν ξέρω αν το βλέπουμε. Γίνεται η μεγαλύτερη νομική, πολιτική, θεσμική αναδριάρθρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι έχει γίνει μέχρι τα, μέχρι τα σήμερα. Και μάλιστα, και αυτό το κίνδυνο το βλέπουν οι εισηγητές προς τιμήν τους, πάει να αλλάξουν οι συνθήκες μέσω κανονισμού. Αυτή λοιπόν η αναδιάρθρωση νομικά και θεσμικά δεν στέκει. Θα είναι τόσο ριζική που αυτό που ξέρουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα θα είναι κάτι διαφορετικό αυτό που θα γίνει αύριο. Και επομένως να τελειώσω με την εξής τώρα, το εξή δίλημα. Χαμένη ευκαιρία με το ότι δεν βγάλαμε σωστά συμπεράσματα ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έκθεση Μπερέζ κρίση, κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Τώρα είμαστε συνυπεύθυνοι. Θα σωθεί η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αυτό το πακέτο ή θα είναι η χαριστική βολή σε αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση και πάμε σε κάτι άλλο. Εύχομαι να μην είναι το δεύτερο. Εύχομαι να μην είναι το δεύτερο. Με αυτή την έννοια λοιπόν η δική μας προσπάθεια είναι στα κείμενα και τις φιλότιμες προσπάθειες των εισηγητών να συμβάλλουμε όσο είναι δυνατόν να γίνουν καλύτερα. Όπου είναι δυνατόν δεν θα αρνηθούμε αυτή την ευθύνη αλλά ταυτόχρονα και ταυτόχρονα να ακουστεί η θέση και η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σα ξαναλέω όμω ότι εδώ η πολιτική ευθύνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αν θα αναλάβει την ευθύνη για τόσο ριζικέ ανατροπέ, όχι προ το καλύτερο, είναι πάρα πολύ σημαντική. Ευχαριστώ πολύ. Oui, mes chers collègues. Εγώ ίσως θα σπάσω τη γενική συνένεση που έχει διαγραφεί και την ε, συνένεση η οποία υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μεταξύ των συντηρητικών και των φιλελευθέρων. Μιλάτε για το να αντιμετωπίσουμε το Συμβούλιο και να τονίσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, αυτά που λέτε συμφωνούν ουσιαστικά με το Συμβούλιο. Συμφωνείτε με το Συμβούλιο να ζητήσουμε μια ισχυροποίηση του, μια αυστηροποίηση μάλλον του Συμφώνου Σταθερότητας. Αυτό που θέλετε να κάνετε τελικά είναι να δημιουργήσετε μια πιο υπερκυκλική πολιτική στον προϋπολογισμό και δεν θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα ελλείμματα της Ευρώπης, θα τα επιδεινώσετε. Θα πνίξετε την ανάπτυξη που ίσα ίσα προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι σήμερα και θα αυξήσετε τα ελλείμματα, γιατί χρειαζόμαστε αντικυκλικές και όχι υπερκυκλικές πολιτικές, αν θέλουμε πραγματικά να τονώσουμε την ανάπτυξη. Δεύτερον, συμφωνείτε με το Συμβούλιο, γιατί θέλετε να δημιουργηθεί ένα δεύτερο υπερσύμφωνο σταθερότητος. Και εδώ μιλάμε για σταθερότητα στις αποδοχές των εργαζομένων. Όταν προτείνεται να υπάρχει προσαρμογή μισθολογική. Προσπαθήστε να σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό. Μας προτείνεται μια κατάσταση η οποία θα αυξήσει ιδιαίτερα την ιδιωτική χρέωση των οικοκυριών που θα χάσουν ε, την ε, αγοραστική του δύναμη και θα δημιουργήσετε μια κατάσταση που θα θυμίζει αυτή της Ισπανίας σήμερα. Και επίσης προσέξτε τις κυρώσεις, γιατί υπάρχει και μια αντιευρωπαϊκή τάση που αναδύεται σε πάρα πολλέ χώρε και επειδή έρχομαι από τη Γαλλία ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει αυτό και θα το δούμε στι επόμενε εκλογέ. Προσοχή λοιπόν στι κυρώσει γιατί διακυβεύεται η ίδια η ευρωπαϊκή ιδέα με όλα αυτά. Τέλο, σε σχέση με την έκθεση τη Vicky Ford, στην οποία είμαι σκιώδη συγητή, πάρα πολλά πράγματα έχουν συζητηθεί. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με το όργανο το οποίο θα ελέγχει την στρατηγική του προπολογισμού των κρατών μελών. Η έκθεση λέει ότι θα είναι ανεξάρτητο αυτό το όργανο. Τι θα πει ανεξάρτητο. Ανεξάρτητο όπως το βλέπει η συγγήτρια. Φαντάζομαι ότι εννοεί ανεξάρτητο από τα κράτη-μέλη. Αν είναι ανεξάρτητο έναντι των κρατών μελών. Δεν μπορεί να είναι ένας ιδιωτικός φορέας όπως οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης που είδαμε ότι τα κάναν θάλασσα, ότι υπερτιμούν ή υποτιμούν τους κινδύνους που συνδέονται με το κρατικό χρέος. Σε αυτήν την περίπτωση λοιπόν θέλουμε να κάνουμε εμείς μία κρίση γιατί υπάρχει ένα τέτοιο ανεξάρτητο όργανο το οποίο ονομάζεται Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και έχει ζητήσει στο παρελθόν η κυρία Μπερέ να μεταβληθεί σε ένα φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και επαναλαμβάνω αυτή την πρόταση. Συγγνώμη που δεν ήμουν απόλυτα πολιτικά ορθός αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή διακυβεύεται το μέλλον της Ευρώπη. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως νομισματική ένωση χωρίς πολιτική ένωση έχει μειονεκτήματα σε καιρό κρίσης. Νομίζω πως ίσως μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτό. Βεβαίω οι απόψει διαφέρουν για το αν πρέπει να έχουμε πολιτική ένωση για να το λύσουμε αυτό το θέμα. Οι έξι αυτές εκθέσεις δεν απαντούν στα μεγάλα ερωτήματα. Το πού πάει η Ευρώπη. διαφωνώ με τον συνάδελφο που λέει πως είναι πολύ εκτεταμένες και βαθιές οι αλλαγές εντός της Ένωσης δεν είναι τόσο βαθίε όσο λένε κάποιοι μιλητέ. Αυτό το οποίο προσπαθούμε πραγματικά να διορθώσουμε, να κάνουμε, είναι να δώσουμε κάποια ουσία στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Όλη η οικονομική ανάλυση των τελευταίων δύο ετών δεν λέει, κανείς δεν έχει πει, πως ε, αυτό δεν είχε καμία σχέση. Το, το υπερβολικό χρέος δεν ήταν πρόβλημα. Και το ότι ακόμα και η Γερμανία και η Γαλλία ξεπέρασαν τα όρια δεν είχε καμία συνέπεια. Όχι. Ε, η συνένεση είναι πως αυτό ήταν μία από τις μεγάλες δυσκολίες που έχει ρίξει την Ευρώπη σε ένα χρέος εμπιστοσύνης που δεν επηρεάζει τα υπόλοιπα μέρη του κόσμου. Οπότε η οικονομική κρίση είναι ήδη αρκετά μεγάλο βάρος και τώρα έχουμε την εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη η οποία φαίνεται πως είναι άμεση συνέπεια της κατάφορης παραβίασης του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Οπότε τι πρέπει να γίνει για να λειτουργήσει αυτό το σύμφωνο. και θεωρώ πως συνολικά η πρόταση της Κομισιόν ε, είναι αρκετά ορθή. Ε, μιλάμε τώρα για μαστίγια και καρότα και δεν χρειαζόμαστε τόσο πολλά μαστίγια και περισσότερα καρότα. Είχαμε αρκετά καρότα, αν θέλετε, στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω πως είχαμε μόνο καρότα. Αλλά δεν είχαμε κανένα μαστίγιο. Και εγώ εκπροσωπώ τη Λετωνία, ένα από τα μικρότερα τη μελη ε, Δεν ξέρω. Και ίσως και από τα πιο. Ίσως όχι από τα πιο περήφανα. Θέλω δεν ξέρω εάν ε, φτάναμε σε μία κατάσταση στην οποία είναι ξέρω η Λετωνία ή η Φιλανδία να έχει παραβιάσει συνθήκες και από την άλλη η Γαλλία και η Γερμανία και να δούμε ποιος θα τιμωρηθεί. Δεν ξέρω εάν το μικρό κράτος μέλος θα μπορούσε να αποτρέψει με τις ψήφους την ε, τιμωρία του. Αλλά το μεγαλύτερο κράτος μέλος, πιέζοντας όλους τους μοχλούς που έχει στη διάθεσή του, θα μπορούσε ίσως να το καταφέρει. Οπότε, για το καλό της Ένωσης, της Ευρωζώνης και χωρών σαν τη δική μου που τώρα έχει μπει στο... έχει προσδέσει το νόμισμά του ευρώ και θέλει να μπει σε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει ένας αυτοματισμός στα μαστίγια. Εάν δεν υπάρχει, αν θέλετε, αυτοματισμός, θα ενθαρρύνουμε κάποια κρατημέλη να συμπεριφερθούν πιθανώς ανεύθυνα, αλλά αυτά τα αρνητικά αποτέλεσμα θα μας επηρεάσουν όλους και τη δική μου χώρα, όπως βλέπουμε σήμερα. Οπότε, συμφωνώ πως χρειαζόμαστε περισσότερα καρότα, νόστιμα τα καρότα κτλ αλλά χρειάζεται και το μαστίγιο. Και το δείχνει αυτό η ιστορία των τελευταιων δυο δύο-τριών ετών. Για να περάσουμε τώρα κατευθείαν στην, στην τέταρτη έκθεση, στην οποία είμαι σκιώδης Υπάρχει ένα ζήτημα οικονομικών προβλέψεων για μια χώρα. Όταν σκεφτόμαστε το προληπτικό χαρακτήρα αυτής της νομοθεσίας, και εδώ πέρα διαφωνώ με κάποιους συναδέλφους που λένε μιλάμε για το μέλλον, εμείς χρειαζόμαστε αυτή την νομοθεσία για να λύσουμε την κρίση σήμερα το απόγευμα. Όχι, η νομοθεσία λειτουργεί συστημικά και μακροπρόθεσμα. Αν είναι καλή νομοθεσία θα προλάβει την επόμενη κρίση. Αλλά αυτή η νομοθεσία, ακόμα και αν εφαρμοστεί πλήρως και με μεγαλύτερα αν θέλετε μαστίγια, δεν είναι αυτή η οποία θα λύσει το πρόβλημα εμπιστοσύνη του σημερινού. Θα βοηθήσει αλλά δεν θα το λύσει από μόνη της. Οπότε, αν κοιτάμε έτσι, μακροπρόθεσμα, την πρόληψη, πρέπει να δούμε σε τι βασίζονται οι προβλέψεις. Και η πρόταση της Κομισιόν ε, ίσως είναι κάπως αντικρούμενη. Γιατί λέει η Κομισιόν, ε, ξέρω εγώ, θα αυξηθεί, θα μειωθεί το ΑΕΠ κατά 100% και θα λέει το κράτος μέλος, όχι τα νούμερά μας είναι διαφορετικά. Θα το συζητάμε αυτό, ποιο έχει δίκιο, ποιο έχει άδικο Νομίζω πιο παραγωγικό θα ήταν η Κομισιόν και κάθε κράτος μέλος να συμφωνήσουν σε έναν αλγόριθμο για το πώς θα βγαίνουν αυτές οι προβλέψεις για να αποφευχθούν πιθανές διαφωνίες. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν οι διαφωνίες, μας ενδιαφέρει η καλύτερη δυνατή ανάλυση ε, για κάθε κράτος μέλος και βεβαίως για την Ένωση. Συνολικά ευχαριστώ. Thank you, Σβέν. Ο Συνάδελφοι, είναι αργά και θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ όλους και όλες που πήραν μέρος σε αυτό το εγχείρημα. Στο πλαίσιο της εποπτείας είδαμε ότι είναι δυνατόν να συνεργαστούμε διακομματικά. Βέβαια, Πολλέ φορέ αυτό δεν συμβαίνει. Σε αυτή την περίπτωση είναι μάλλον ακριβώς αυτό. Δηλαδή είναι δύσκολο γιατί οι πολιτικές διαφορές είναι μεγάλες. Από την άλλη μεριά οι πολίτε παρακολουθούν πολύ προσεκτικά τι θα κάνουν αυτή τη στιγμή και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε όσο πιο πολύ γίνεται να καταλήξουμε σε κάτι που να είναι λειτουργικό, οικονομικά και ταυτόχρονα είναι δίκαιο γιατί αυτά τα δύο τα παρακολουθούν οι πολίτες με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πολλοί συνάδελφοι ανάφεραν ότι το προτινόμενο πακέτο της Κομισιόν έχει μόνο μερικά στοιχεία για μια αναγκαία λύση. Είναι τυφλό από κάποια σκοπιά και πρότεινε και συμφωνώ με την συνάδελφο που το είπε προτείνει και ορισμένα περιτά πράγματα. Ναι, να υπάρξει σταθερότητα, να ενισχυθεί η σταθερότητα. Από την άλλη μεριά όμως, αν δούμε μόνο τις δαπάνες, το σκέλος δαπάνη, καταστρέφοντας συστηματικά την ικανότητα κρατών μελών να αυξήσουν τα φορολογικά τους έσοδα δεν αρκεί. Ένα δεύτερο θέμα, κομβικό, πρέπει να είναι σαφές ότι αν υπάρχουν ανισομέρειες, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πλεονάσματα και ελλείμματα. Αυτά πάνε πακέτο. Πρέπει να κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά ποιο δημιουργεί τι. Όχι να πούμε όποιο είναι σε έλλειμμα είναι ένοχος πάντα και όποιο έχει πλεόνασμα πάντα πρέπει να είναι το αφεντικό και ο πιο καλός. Ελπίζω να είμαι σαφής σε αυτά που λέω. Τέλος, η κατάσταση εδώ που συζητάμε δεν συζητάμε εν κενό. Συγκεκριμένες χώρες υποφέρουν από την υποχρέωση. Ακόμα και η πιο πλούσια χώρα. Κάποιος αναφέρθηκε στη Γερμανία, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες. Και αυτές θα πρέπει να κρίνουν. Τελικά είναι πιο φθηνό να ανοίξει η συζήτηση για την πραγματική φορολογική συνεργασία πρόσβαση σε κεφάλαια ή ακόμα και αναδιάρθρωση του χρέους ή απλή διαγραφή του χρέους χωρίς τα μέτρα που ανάφερα πριν. Θεωρώ λοιπόν ότι το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να χρησιμοποιήσει την τρέχουσα συγκυρία να επιμείνουμε σε κάτι που είναι λειτουργικό και όχι να περιοριστούμε σε πολύ τεχνικές λύσεις η Σάμφος Γκούλαρ με αυτό που πρότεινε διευρύνει το πλαίσιο και νομίζω ότι οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις οχρές κοιλίδες όπου υπάρχουν. Και συμφωνώ με τους συναδέλφους που επεσήμαναν ότι ένας απλός αυτοματισμός δεν αρκεί. Χρειαζόμαστε την ικανότητα να κινηθούμε προς μια πραγματική οικονομική ένωση που θα μπορεί να παίρνει αποφάσεις που θα έχει τα όργανα που χρειάζονται για να παίρνει τεκμηριωμένες αποφάσεις, τουλάχιστον στην Ευρωζώνη, και αυτό το πλαίσιο είναι στο κοινό συμφέρον του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να είναι η κοινοτική μέθοδος, όχι η μέθοδος του Συμβουλίου. Η κοινοτική μέθοδος πρέπει να διέπειτα τα της Ευρωζώνης και ελπίζω να εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με αυτό το πνεύμα. Και είμαι, και σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή η πραγματικότητα, τα, τα, τα καθαρά οικονομικά νούμερα θα κινήσουν τη συζήτηση προς την κατεύθυνση αυτή. Το απλώς να αναμορφώσουμε το σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και να επιμένουμε στην σταθερότητα δεν θα μας βγάλει από την κρίση. Η πραγματικότητα θα οδηγεί στην συζήτηση προς την κατεύθυνση που είπα. Πρόεδρος, τέσσερι ακόμη συνάδελφοι έχουν μείνει να μιλήσουμε. Δύο λεπτά παρακαλώ ο καθένας. Mark. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω να πω καταρχήν ότι συμφωνώ πάρα πολύ με αυτά που είπε ο κ. Κάρινς εδώ. Είναι δύο πράγματα ακόμα τα οποία πρέπει να πω για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτό το. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το, αυτά τα νομοθετήματα. Γιατί σε μια σύγχρονη οικονομία όλα συνδέονται. Το πόσο επενδύουμε έχει να κάνει με την μελλοντική ανάπτυξη και με την οικονομική σταθερότητα. Αλλά επίσης το τι κάνουμε για την εκπαίδευση, τι κάνουμε για την παιδική φροντίδα κτλ. Και μπαίνουμε πια σε μια πραγματική πολιτική συζήτηση. Και εδώ δεν μπορούμε να έχουμε τον πραγματικό έλεγχο για τα εργαλεία τα οποία εξασφαλίζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα. Και η συζήτηση που κάνουμε σήμερα εδώ μας το υπενθυμίζει. Εγώ νομίζω ότι ένα από τα πιο σημαντικά είναι να, <clears throat> πράγματα είναι να εστιάσουμε στα κριτήρια του βαθμολόγιου που έχουν πραγματικό ουσιαστικό αντίκτυπο στην δημοσιονομική σταθερότητα, στην χρηματοοικονομική σταθερότητα, που είναι τα πλεονάσματα και τα ελλείμματα, το ισοζύγιο τρέχουσών συναλλαγών. Υπάρχουν κάποιες μακροοικονομικές ανισομέρειες που είναι Κεφαλαιόδηση. Θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας εκεί. Γιατί βλέπω να υπάρχει μια τάση να πολλαπλασιάσουμε τα βαθμολόγια και να κάνουμε τη συζήτηση αυτή πολιτική. Όσο περισσότερα κριτήρια έχουμε, τόσο λιγότερο σημαντικό θα είναι το κάθε, από τα, σημαντικό το κάθε κριτήριο και περισσότερη πολιτική συζήτηση θα έχουμε για την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας. Η δεύτερη παρατήρησή μου είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι να μην αντιμετωπίσουμε μονάχα τα ελίματα αλλά και τα πλεονάσματα στις εποχές παχαίων αγελάδων. Και πρέπει να ενισχύσουμε τους στόχους μας ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τα πλεονάσματα αυτά. Όχι μονάχα να υπάρχει μια συζήτηση για το πόσο αξιόπιστη είναι η προβλέψεις των κρατών μελών. Γιατί κάθε χώρα έχει το κάθε συμφέρον να είναι αξιόπιστη. Και δεν μπορεί κανείς να φαντάσει ότι η Κομισιόν μπορεί να μετράει καλύτερα από τα κράτη-μέλη, αλλά θα πρέπει να παρακολουθούνται οι η επίτευξη των στόχων για το πόσο σε μια μακρύτερη χρονική περίοδο μπορεί ένα κράτο να εξασφαλίσει την ισορροπία των δημοσιονομικών. Έχω και άλλα πράγματα να πω, αλλά δεν προφέρω να τα πω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρο. Ο Λάιος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μόνο μία. μόνο παρατήρηση, γιατί ήρθε ο ξανά και ζήτησε συμβουλή για την τροπολογία αυτή, 27 για το 1 20 και νομίζω πως και οι δύο επιλογές είναι κακές. Αν θέλετε την ταπεινή μου γνώμη, δεν μπορούν να λειτουργήσουν στην πράξη. Αν κάνετε ένα απλό υπολογισμό, βλέπετε πως στην περίπτωση της χώρας σας εξαρτάται από τις υποθέσεις που έχουν γίνει, δηλαδή πως η ανάπτυξη και προπολογισμό προβλέπει κανείς και την φύση της χρηματοδότησης του χρέους. Οπότε εδώ πέρα έχουμε το πρόβλημα του αποθέματος και του χρέους. Αν υπάρχει μια χώρα σαν την Ελλάδα με χρέος 135% του ΑΕΠ είναι απελπιστική η κατάσταση. Αν έχουμε μια χώρα με μόνο 70% ε, μπορεί να, να λειτουργήσει και να έχει νόημα, αλλά μόνο αν έχουμε ανάπτυξη. Αν δεν έχουμε, έχουμε το ίδιο πρόβλημα όπως ε, ανέφεραν πάρα πολύ συνάδελφοι εάν θέλουμε δηλαδή να έχουμε μια αντικυκλική φιλοκυκλική πολιτική και κάποιο ε, κάποιος δεν χρησιμοποίησε τον καιρό των παχιών αγελάδων για να συσσωρεύσει πλεονάσματα, τότε δεν έχει επιλογή παρά να ακολουθήσει μια φιλοκυκλική πολιτική. Όσοι είχαν δε το προπατορικό αρμάρτημα τον καλό καιρό να ξοδεύουν, έχουν σήμερα την τιμωρία του να μην μπορούν να ακολουθήσουν αντικυκλικές πολιτικές τους δύσκολους καιρούς. Οπότε πρέπει να διαχωρίσουμε από θέματα προές, πρέπει να δούμε την αφετηρία όπως σας είπα, το προπατορικό αμάρτημα και την ροή του πώς θα φτάσουμε σε κάτι πιο βιώσιμο από ε, οικονομική σκοπιά. Ευχαριστώ πολύ, σας. Ευχαριστώ. Θα θεμεγήσω όσες εισηγήτρια της Επιτροπής Απασχόλησης για τρεις από τις έξι εκθέσεις της κυρίας Βόρτμαν Κόλ, της κυρίας Φερέρα και του κυρίου Χάντλουντ. Και σας θυμίζω ότι στο πακέτο αυτό θα παραμείνουν μερικά απομεινάρια leftover της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Αυτά τα υπόλοιπα, τα απομεινάρια θα πρέπει να μας βοηθήσουν στη συζήτηση που κάνουμε. Γιατί όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση κάναμε σαν αυτό που γίνεται στο Συμβούλιο να μην έχει σημασία. Α, μια απλή, μια απλή αναθεώρηση που θα αφορά τα βασικά σημεία, σημαντικά σημεία που είχαμε αναφέρει εμείς στην έκθεση της Επιτροπής της Κρίσης που ελπίζω να έχετε την ευκαιρία να ε, συζητήσετε και να αποφανθείτε γι' αυτό όταν θα έρθουμε στο θέμα της αναθεώρησης της συνθήκης. Τηλεγραφικά και λακωνικά για το τι προτείνω εγώ στην Επιτροπή Απασχόλησης. Πρώτον, μας ανησυχεί κάπως μια ποσοτική προσέγγιση, ενώ το σύμφωνο σταθερότητα απέδειξε ότι είναι ανίκανο για δράση σε τέτοια θέματα, στη μείωση των αποκλήσεων ανταγωνιστικών, στην ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών. Η τραγωδία του Συμφώνου Σταθερότητας είναι αυτή ότι θα έπρεπε να επιτρέψει σε χώρες που έχουν διαφορετικές συνθήκες να ζουν με το ίδιο νόμισμα. Τι είδαμε, μια ποσοτική μόνο προσέγγιση που οδήγησε σε απόκληση στο βαθμό ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών αυτών. Δεύτερον, στο θέμα της prudent fiscal policy, να το αντικαταστήσουμε με την εξίσου δύσκολη έννοια του efficient fiscal policy, αποτελεσματική, αποδοτική δημοσιονομική πολιτική. Γιατί με τις γενικές δημογραφικές ανισομέρειες που βλέπουμε και τις τεράστιες παγκόσμιες προκλήσεις έχουμε κάθε λόγο να θέλουμε να προχωρήσουμε θετικά προς το μέλλον. Τρίτο, το σύνολο του πακέτου που προτείνει η Κομισιόν στηρίζεται μόνο στο άρθρο 121 της Συνθήκης, η οικονομική πολιτική. Για άλλη μια φορά τα θέματα απασχόλησης βλέπουμε τι χειρισμό έχουν. Βάσει το άρθρο 148 η Ένωση έχει ευθύνη έναν των κρατών μελών και για τα θέματα αυτά. Σας καλώ λοιπόν να δείτε κατά ποιους όρους και συνθήκες είναι δυνατόν το σύνολο του πακέτου να στηρίζει στην διπλή αυτή νομική βάση και το 121 και το άρθρο 148 να μην έχει αυτή την ε, ε, μεταχείριση ως μια απλή παράμετρο στο θέμα της απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε την Περβάνς. Άστριντ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξαναγυρίσω στα προηγούμενα της χρηματοοικονομικής εποπτείας. Ήταν ένα σφάκελος όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο γιατί μπόρεσε να έχει ένα πιο ευρωπαϊκό και συνεκτικό τρόπο αντιμετώπιση. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να παίξει και στο τρέχον ζήτημα ένα αντίστοιχο ρόλο, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε απόλυτη ε, επίγνωση του ότι περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερη ε, αυστηρότητα. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα διαλύσουμε όλα στο όνομα της λιτότητος και της πειθαρχίας, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε περισσότερη ευρωπαϊκή ενοποίηση και συγχρόνως να μην υποστηρίζουμε τις αρχές της χρηστής διαχείρισης του προϋπολογισμού. Ε, κάποια πράγματα για τα ευρωομόλογα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να μιλήσουν καθόλου για αυτά. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, γιατί υπάρχει σύγχυση αυτή τη στιγμή στη συζήτηση. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ακριβώς γιατί μιλάμε για τα ευρωομόλογα. Αυτό εξαρτάται από τη μορφή των ευρωομολόγων που θα επιλέξουμε και οι συνέπειες από τις επιλογές αυτές είναι σημαντικές. Πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε για τα θέματα αυτά, αλλά έχω και ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Για να καθορίσουμε τα κριτήρια του δημόσιου ελλείμματος του 3% μέχρι στιγμής, αυτό ελάμβανε υπόψη τη δημοσία διοίκηση, και την, ε, τις παροχές κοινωνικής ασφάλειας λοιπά. Βλέπω τώρα ότι θέλετε να βγάλουμε από το παιχνίδι την κοινωνική ασφάλιση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Λουξεμβούργο. 12,7 δισεκατομμύρια είναι ο προπολογισμό του του 2011. 1,2 είναι το έλλειμμα του τα 100 του ΑΕΠ είναι το έλλειμμα της ε, δημόσιας της κεντρικής αλλά συνολικό έλλειμμα της διοίκησης είναι 3%. 1,2 μονάχα στη δημόσια διοίκηση, γιατί είμαστε εξαιρετικά υγιείς και έχουμε ένα υγιέστατο συνταξιοδοτικό σύστημα, τουλάχιστον προς το παρόν. Μα αυτό είναι πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω. επειδή έχουμε ένα αποθεματικό πάνω από 10 δισεκατομμύρια στο δημόσιο συνταξιδοτικό σύστημα, 800 εκατομμύρια πλεόνασμα τα τελευταία χρόνια είχαμε, φτάνουμε σε ένα συνολικό έλλειμμα 1,5% ενώ η δίκηση είναι στα 3,4%. Σας δίνω τους αριθμούς για να σας τα εξηγήσω ο κύριος Γιούνκερ δεν θα χαρεί καθόλου αν βγάλετε τις, ε, τα στεξοδικά ταμεία από τα, από τα κριτήρια. Πρέπει να λάβουμε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία γιατί και ο κρατικός προϋπολογισμός έχει 36% δαπάνες κοινωνικών μεταφορών κοινωνικού χαρακτήρα, 20% μισθοδοσία και 13% επενδύσεις. Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, αλλά σε μεθοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και συγχωρήστε με κυρία Μπερές. Θα έχετε το καιρό ως Επιτροπή Απασχολήσεως που είσαστε συγγήτρια για τρεις εκθέσεις να πείτε ό,τι θέλετε. Οπότε αφήστε να μιλήσουν και τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων και πρέπει να το σκεφτείτε αυτό, να το έχετε στο μυαλό σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκοζές πάρα πολύ σύντομο κύριε Πρόεδρε. Η Αστή δεν μίλησε για την εποπτεία. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο παίζουν κάποιο ρόλο αυτοί οι εποπτικοί φορείς, έτσι όπως θεσπίζονται, πρέπει να προσέξουμε γιατί θα πρέπει να επανέλθουμε στο θέμα αυτό με την ε, μορφή με την οποία θεσπίζονται αυτοί οι φορείς μπορούν να καταστρέψουν όλα αυτά τα οποία πέτυχε το Κοινοβούλιο. Έχω τώρα μια συνάντηση με τη Βελική Προεδρία για να μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Κλείνω τη συζήτηση και σα λέω ότι η οριακή ημερομηνία για τι τροπολογίε είναι η 10η Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Οι εξετάσει των τροπολογιών 21-22 Μαρτίου. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μα 19-20 Απριλίου ώστε να περάσουμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο του 2011. Όλα αυτά είναι ακόμα ενδεικτικά γιατί περιμένουμε τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ και θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί.